Dear colleagues, we will begin today's meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Ο πρόεδρος μας, κύριος Μακάλιστερ, αναγκάστηκε να επιστρέψει για να ε, παραστήσει την κηδεία του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος της Γερμανίας. Εγώ θα προεδρεύσω λοιπόν σχέδιο ημερήσια διάταξη, έγκριση αυτή. Αν δεν διαφωνείτε, έχετε σχόλια, εγκρίνεται. Δεύτερον, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 27-28 Φεβρουαρίου 2017. Αν δεν έχετε σχόλια, θεωρούνται εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Προχωρούμε με ρογούς ρυθμούς. Τρία ανακοινώσει του Πρόεδρου. Με ενημερώνει η γραμματεία ότι δεν έχω ανακοινώσει να σας κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε και θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 4. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών. Τέσσερα, πάρα πολύ σημαντικό σημείο σήμερα, η έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία του 2016. Είναι μια πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης, πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ επίκαιρη. Όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα στη Μήνη Ολομέλεια, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Τουρκία και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Από πέρσι η Τουρκία ε, γνώρισε μια απόπειρα πραξικοπήματος και πευλήθη στη συνέχεια ε, ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουμε δει και ε, διάφορες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. 16 Τετάρτου έγινε δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του συντάγματος που μπορεί να έχει κρίσιμες επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις ε, σύνδεσης. Η Επιτροπή της Βενετίας έχει εκφράσει αμφιβολίες για το είδο του καθεστώτος που θα επιβληθεί αυτή τη στιγμή αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Την περασμένη εβδομάδα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης ε, ψήφισε μια απόφαση, ένα ψήφισμα για να ξαναρχίσει η παρακολούθηση ε, της Τουρκίας. Ε, εμείς ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Χάν να καλεί ε, για να δούμε ένα νέο τύπο σχέσεων με την Τουρκία αφού εμεί στο παρελθόν είχαμε ζητήσει ε, και ψηφίσαμε να παγώσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσει. Και έρχεται η έκθεση αυτή να συνεισφέρει στην όλη ε, περισυλλογή και στον προβληματισμό μα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να στείλουμε αποστολή τις ερχόμενες εβδομάδες της Επιτροπής μας μαζί με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Άγκυρα. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Πύρη, Θυμίζω ότι η προθεσμία απολογιων τροπολογιών είναι 9η Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Κυρία Πύρη, έχετε το λόγο, this Ελπίζω να σας βλέπουμε πιο συχνά, Πρόεδρε, γιατί πράγματι προχωράτε πολύ αποτελεσματικά και γρήγορα. Λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι εδώ γιατί χθε ήταν γιορτή, ιδιαίτερα για τους Κυπρίους ήταν μακριά, δεν ήταν εύκολο λόγω της ε, εορτής να βρει κανείς πτήσεις. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση της κατάθεσης της έκθεσης. Αυτό οφείλεται στο δημοψήφισμα που έγινε στην Τουρκία έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία απόφαση πριν από τις διακοπές για το πώς βλέπουμε τις σχέσεις με την Τουρκία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το 2016 για τον τουρκικό λαό ήταν ένα άνους ορίμπιλης προβλήματα με τον πόλεμο στη Συρία, τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, και φυσικά μια ολόκληρη σειρά τρομοκρατικών επιθώσεων με αποκορύφωση φυσικά και το πραξικόπημα. Το μόνιμο πλέον καθεστώς έκτακτης ανάγκης διασφαλίζει ότι ότι για τους 140.000 απολυθέντες και τις 14.000 ε, που έχουν κρατηθεί ή φυλακιστεί κατά καιρού, δεν έχουν καμία δυνατότητα μέσω των τακτικών διαδικασιών να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους. Είδαμε τη φυλάκιση επίσης όχι μόνο δημοσιογράφων αλλά και συναδέλφων κοινοβουλευτικών προημερών ε, φυλακίστηκαν άλλοι 13 ε, βουλευτές μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνο του κόμματός τους ο κύριος Ντεμιρτάς. Ε, πάρα πολύ πανεπιστημιακή, περισσότεροι πανεπιστημιακοί παρά στρατιωτικοί εν πολλής, και αυτό είναι λίγο περίεργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει επίσης ε, συστηματικά ε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανεξαρτησία και του τύπου και του δικαστικού. Το 1 πέμπτο των δικαστών και των εισαγγελέων απελήθησαν και υπάρχουν και επιμέρους νομικές ρυθμίσεις οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν την επιρροή μέσω της Άγκυρας και της τουρκικής διασποράς του προβλήματος της Τουρκίας στις χώρες μας. Αν δούμε την λεπτομέρεια, το μέγεθος και την σοβαρότητα των τουρκικών αρχών σαν παράδειγμα παρακολούθηση των μελών της τουρκικής διασποράς της αντιπολίτευσης από τις ημιστικές ε, υπηρεσίες όπως επίσης ε, και εκφοβισμοί μελών της διασποράς. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να θέσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην το περιορίσουμε σε διμερές κατά περίπτωση. Για το δημοψήφισμα τώρα, παρά το ότι το σύστημα το εκλογικό ήταν άδικο και ανελεύθερο εν πολλής, έχουμε αμφιβολίες επί το, επ' αυτού δηλαδή, οι μισοί σχεδόν Τούρκοι ψήφισαν υπέρ της δημοκρατίας της χώρας τους. Αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία στην Τουρκία δεν έχει αποθάνει. Εκατομμύρια Τούρκοι όμως ψήφισαν υπέρ μιας πρότασης η οποία θα απομακρύνει την Τουρκία από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ο παράγων φόβος έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση αντέδρασε και είναι θετική και η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είπε ότι εφόσον δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις εξουσίες είναι σαφές ότι η Τουρκία αποκλίνει των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Το Νοέμβριο ε, το κοινοβούλιο μας με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε να παγώσει προσωρινά την διαδικασία ένταξης ελπίζοντας ότι η χώρα θα επέστρεφε σε δημοκρατικές αλλαγές. Δυστυχώς όμως το καθεστώς έκτακτης ανάγκης παραμένει και βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει από τον μήνα Νοέμβριο και στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συστηματική παραβίαση των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Αυτό θα οδηγήσει σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπενχάγης ακριβώς και στην διακοπή των διαπραγματεύσεων. Και αυτό είναι αυτό το οποίο λέγω και στην πρότασή μου, αλλά θέλω να ακούσω και τις απόψεις σας. Εγώ δεν διεκδικώ ε, το να κλείσουμε την πόρτα στην Τουρκία ή να σταματήσουμε πλήρως τη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Ε, είναι δύσκολες οι σχέσεις βέβαια με την Τουρκία και θα γίνουν ε, πιο δύσκολες αν ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίσει τη ρητορική που ακολούθησε τις τελευταίες εβδομάδες για την ναζιστική Ευρώπη, την ναζιστική Γερμανία κτλ αλλά με ένα τέτοιο νέο σύνταγμα είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι λοιπόν η δυνατότητα μόχλευσης την οποία έχουμε. Ε, δεν παίζει πια αν θέλετε το, το, η διαδικασία, το δόλωμα της ε, ξεκίνησαν μεταρρυθμιστικές ε, διαδικασίες ήδη από το 2004, παρόλα αυτά ίσως και δεν κάναμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Εμείς ζητάμε να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24 εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν συνέβη ποτέ αυτό. Τίθεται επίσης ε, και προβλήματα για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται να αμφισβητήσει η δική μας αξιοπιστία όταν βλέπουμε το τι συμβαίνει σε χώρες όπως η Ουγγαρία. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης, δεν είναι μόνο για μας σημαντικό αλλά και για την ίδια την Τουρκία η οποία περνά δύσκολους οικονομικούς καιρούς αλλά μόνο εάν συνοδεύεται από ξεκάθαρα, αν θέλετε, ξεκάθαρος ε, ε, δίκτες που θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Τώρα να μιλήσω λίγο για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν το καλοκαίρι. Είναι καλό που θα γίνει στις 25 Μαΐου μια συνάντηση κορυφής, μια μίνι συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν θα είναι εύκολα. Είναι καλό επίσης ότι ε, προσκλήθηκε ο Πρωθυπουργό στη Μάλτα. Αλλά η αντίδραση της τουρκικής πλευράς σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στη Μάλτα μας δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία. Ε, και μάλιστα άλλοι 4.000 ε, ε, ξεδιώχθησαν από τις θέσεις τους μετά τις συζητήσεις αυτές και ταυτόχρονα αποκλείστηκε η πρόσβαση και στο, στην ιστοσελίδα της Wikipedia. Η Επιτροπή είπε μετά το, <clears throat> το δημοψήφισμα ότι θα υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Ε, τώρα πια δεν γίνεται ούτε καν αναφορά στις παρατηρήσεις της ανεξάρτητης ομάδας εποπτείας της, ε, του ε, ΟΑΣΕ. Η κυρία Μογκερίνη μετά από τη δημοσίευση της Επιτροπής της Βενετίας είπε ότι θα αξιολογήσουμε το πώς το νέο συνταγματικό πακέτο, αν θέλετε, ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ε, για το 2018. Εγώ νομίζω ότι το πακέτο των, δημοκρα... των ε, συνταγματικών αλλαγών είναι δεδομένο και γνωστό. Οι αξιολογήσεις της ευρωπαϊκής πλευράς είναι σαφείς, οπότε γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2018. Και τι γίνεται με το μήνυμα που στέλνουμε στα εκατομμύρια των Τούρκων που παλεύουν για την δημοκρατία στη χώρα αυτή τους λέμε ότι κοιτάξτε εμείς θέλουμε κάποιες ε, διαπραγματεύσεις ε, οι οποίες ε, θα είναι διαμεσολαβητικές ίσως αλλά δεν θα πρέπει να θίξουν τα πολλαπλά μας οικονομικά κριτήρια. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι μελλοντικές σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξουμε οδήποτε κόστος θα πρέπει να ζητήσουν ξεκάθαρες φωνές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση των δημοσιογράφων, την απελευθέρωση του Ντέμιρτας, να τεθεί τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια τελική παρατήρηση. Ξέρω ότι υπάρχουν μεταξύ μας πάρα πολλές διαφορές. Οι διαφορές αυτές σοβούν ήδη από το 2004 ε, βλέπουμε τις σχέσεις με την Τουρκία με διαφορετικό τρόπο. Ο μοναδικός τρόπος όμως με τον οποίο μπορούμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην συνάντηση του Συμβουλίου τον Ιούνιο είναι να είμαστε ενωμένοι. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι για τον μισό τουρκικό πληθυσμό που δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωση της δημοκρατίας στην χώρα αυτή και εμείς θα πρέπει καθημερινά να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να μην λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα σε εισαγωγικά ε, στην χώρα αυτή. Πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο σαν κοινοβούλιο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλούς από μας και γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο σε όλους τους σκιώδεις για 3,5 λεπτά στον καθένα. Ιωσδήποτε άλλος θα ήθελε το λόγο θα πρέπει να το δηλώσει αυτό όσο μιλούν οι σκιώδεις. Και θα προσπαθήσουμε αφού έχουμε κλείσει τον κατάλογο να μοιράσουμε τον χρόνο για να μπορέσουν όλοι να πάρουν τον λόγο. Λοιπόν, πείτε μου ποιος θέλει το λόγο κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Θα ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Ζωμά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ αυστηρός είστε σήμερα. Ε, θέλω να, ζητήσω, να ευχαριστήσω μάλλον τη συνάδελφο Κάτι Πύρη για το σχέδιο έκθεσής της και για τα σταρά τα λόγια που μας είπε. Και ε, την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέρη επίσης τοποθετήθηκε αντίστοιχα. Είναι λίγο δύσκολο να βρούμε απαντήσεις με το ψήφισμα αυτό στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Τουρκία, γιατί από τον Οκτώβριο έχουν γίνει πάρα πολλά από τότε που εκδόθηκε η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουσιαστικά θα κάνουμε εμείς έκθεση της κατάστασης για την Τουρκία, όχι Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα πίστευε Και όποιο νόμιζε πριν από λίγε εβδομάδε ή μήνες ότι έχουμε δει τα χειρότερα, εξεπλάγει. Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο στη σχέση μας με την Τουρκία και θέλω να υπογραμμίσω ότι βεβαίως είναι σημαντικές οι σχέσεις. Πρέπει να έχουμε σχέση με την Τουρκία, είναι άμεσος γείτονας όσο και σημαντικός. Εμπορικός εταίρος, σημαντικός επαναλαμβάνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να διακόψουμε τις σχέσεις μας και τις ε, συνεργασίες. Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν το καθεστώς υποψήφιας χώρας είναι το σωστό ε, πλαίσιο για να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε και σωστά το κάνουμε τι θα κάνουμε στη σχέση μας με αυτή τη χώρα. Και η Επιτροπή Βενετίας βεβαίως διαπίστωσε ότι η αναθεώρηση του συντάγματος που πέρασε με μικρή διαφορά στο δημοψήφισμα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που εμείς θεωρούμε δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αν γίνει πραγματικότητα αυτό το καθεστώς που προβλέπει λοιπόν η αναθεώρηση του συντάγματος, με τον τρόπο που προτείνεται, χωρίς την παραμικρή αλλαγή, τότε θα έχει έρθει η ώρα να πούμε ότι φτάνει πια. Αυτή είναι κόκκινη γραμμή επέναντι στην Τουρκία. Τώρα, και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Το να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις, να παγώσει όλο το ζήτημα ε, επαόριστο ή να τερματιστεί το καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις εκταμιεύσει προς την Τουρκία αν δεν διακοπούν οι διαπραγματεύσεις. Και μέχρι πότε θα παγώνουν οι διαπραγματεύσεις και θα αναβάλλονται δεκαετίες, πόσο θα κρατήσει αυτό μετά τη συνταγματική ενθεώρηση. Είναι διαβίου πρόεδρος είναι πρόεδρος της Τουρκίας και θα κυβερνάει όπως θέλει και θα εξακολουθούμε εμείς να δίνουμε λεφτά στην Τουρκία. Αυτό δεν μπορώ να το πω σε κανένα πολίτη στη χώρα μου. Γενικά μου αρέσει το σχέδιο έκθεση τη εισηγήτριας, μου λείπουν όμω μερικά σημαντικά σε κρίσιμα σημεία και στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσα συζητήσαμε πέρυσι. Για την Κύπρο θα πρέπει να πούμε πολύ περισσότερα και έχω απογοητευτεί αγαπητή κάτι που δεν τα έχεις ξανά όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει ε, και ε, τα περισμένα χρόνια και πέρυσι βάλαμε μετά από διαπραγματεύσεις το κείμενο. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Θα ήθελα και κάτι για την ε, ανεξιθρησκεία και την ελευθερία της θρησκείας που διακυβεύεται και απειλείται όλο και περισσότερο στην Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Μπέλντερ από την ομάδα ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ACR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πύρη, με ε, ενδιαφέρον και ικανοποίηση βλέπω την έκθεσή σας. Στην παράγραφο 4 λέτε ότι δεν συνάδουν με τα κριτήρια της Κοπενχάγης αναθεώρηση του συντάγματος. Και από το 1999 είναι προαπαιτούμενο και προϋπόθεση για την ένταξη μιας χώρας αυτά τα κριτήρια. Λέτε ότι η Τουρκία απομακρύθηκε έτσι περαιτέρω από τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Και σας ερωτώ, θα δώσουμε μια σαφή ευρωπαϊκή απάντηση γιατί χρειάζεται κάτι να πούμε στη Μάλτα έγιναν συζητήσεις και ε, στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung υπήρξε ένα άρθρο και λέτε σε περίπτωση που γίνει αναθεώρηση του συντάγματος να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν δεν απατώμε, και το 2019 Ε, έχουμε νέε προεδρικές εκλογέ. Γιατί έχετε διατυπώσει έτσι αυτή την παράγραφο, δεν το καταλαβαίνω. Στην παράγραφο 8 μιλάτε για τη σοβαρή παραβίαση της ελευθεροτυπίας. Ε, είμαι σε επαφή με δημοσιογράφους και από τη Γερμανία και από τη Τουρκία. Δεν θέλω να σας αναφέρω έντυπο για λόγω ασφαλείας και μίντια. Ε, παρεμποδίζονται οι δημοσιογράφοι να ασκούν το επάγγελμά τους στη χώρα αυτή και δεν μπορούν και να ενημερώνουν σωστά τους πολίτες. Στη Frankfurter Allgemeine επίσης ε, δημοσιεύεται ένα άρθρο πάρα πολύ εύστοχο και έγκυρο. Συμφωνώ με την κυρία Σόμερ. Στην παράγραφο 11 ελπίζω να κάνω και μια τροπολογία σχετικά για την παραβίαση της ε, ελευθερίας της λατρείας και Υπάρχει και μια διαμαρτυρία της Ένωσης Προτεσταντικών Εκκλησιών και επίση λέτε για τον τρόπο με τον επηρεάζει η κυβέρνηση της Τουρκίας και το καθεστώς στη διασπορά τους Τούρκους που ζουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι σημερινό θέμα. Είναι ένα θέμα ετών. Ξέρετε τι γίνεται με το Διανέτ και πώς χρηματοδοτείται από το τουρκικό κράτος. Που είναι το, το Συμβουλίο για ε, θρησκευτικά ζητήματα ε, και έχει πολλές διασυνδέσεις και πολλά πλοκάμια σε διάφορα υπουργεία και το μακρύ χέρι στην Ευρώπη. Στην έκθεσή σας θα πρέπει να διατρανώσουμε ότι έχει χειραγωγήσει πλήρως ο Ερντοάν. Τώρα έχει ε, ε, ε, εξαπολύσει και μια εκστρατεία της Ημισελήνου κατά του Σταυρού και των θρησκευτικών συμβόλων. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Θα κάνω και τροπολογίες. Και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ίσης. Και τέλος, εμείς έχουμε οικονομική επιρροή και θα πρέπει να την ασκήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε. Έχουμε μοχλούς πίεσης για την τουρκική οικονομία. Και αυτά τα λένε και διάφοροι εμπειρογνώμονε και στη Γερμανία ένα πολύ έγκυρο που ασχολείται με τα τουρκικά θέματα, ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοχλό των οικονομικό θα χάσουμε το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Και σα ευχαριστώ και για τη γενοδορία σα το χρόνο. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο αυστηρό λοιπόν. Ο κύριο Λάμστορφ από του Φιλελευθέρου για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και με χαρά βλέπω ότι είστε γενναιόδωρο ω προ τον χρόνο. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω την Κάτι Συμφωνούμε με την παρουσίαση και την περιγραφή της κατάστασης, ε, όπως την αναφέρει η έκθεσή της και μας τα είπε και η ίδια σήμερα προφορικά. Συνεχίζονται οι παραβιάσεις των κριτηριών της Κοπενχάγης. Άρα δεν βρισκόμαστε εμεί σε νομικό κενό ω κοινοβούλιο και είναι σημαντικό αυτό. Ε, όταν λέμε ότι θα πρέπει να παγώσουν, να αναβληθούν, να τερματιστούν οι διαπραγματεύσει, αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σε ένα ε, κείμενο νομικά δεσμευτικό. Δεν πρόκειται εδώ για άγρια πολιτική σπέκουλα και εικασίε. Υπάρχουν αυτά σε ένα θεσμικό πλαίσιο νομοθετημένα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμεί είμαστε το πρώτο θεσμικό όργανο που από πέρσι ζητήσαμε να παγώσουν οι διαπραγματεύσει και συμφωνώ απολύτως με τη συντριβή και ε, την απογοήτευση για την ε, πολύ ασθενή ε, στάση των Υπουργών Εξωτερικών στη συνεδρία Συγκύμνη στη Μάλτα. Μόνο η Αυστρία και το Λουξεμβούργο νομίζω, ύψεσαν τη φωνή τους. Ο Ζίγμερ Γκάμπριελ θεωρεί ότι εντάξει, μπορεί να είναι ακόμα υποψήφια προς ένταξη η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό με ξεπερνάει. Ε, τώρα, θα πρέπει να παγώσει η διαδικασία, θα πρέπει να τερματιστεί. Ε, το ερώτημα αυτό είναι εύλογο. Αλλά από τη σκοπιά τη δική μας, της πολιτικής μας ομάδας, αλλά και άλλων συναδέλφων, ε, θα πρέπει να προτείνουμε κάτι νέο, μια αντικατάσταση. Το θέμα δεν είναι να τερματιστεί ο διάλογος, να γυρίσουμε την πλάτη στην Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις επαφές, το διάλογο και τη συνεργασία, διότι η Τουρκία είναι και θα παραμείνει ένας σημαντικός εταίρος και γείτονας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περήφανος λαός με μεγάλη ιστορία. Έχουμε εκατομμύρια ε, πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουρκικής ε, καταγωγής και μην ξεχνάμε ότι είναι και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ σε μια δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση και είναι προς το συμφέρον της Δυτικής Συμμαχίας η δράση της και δρά υπέρ της ε, Δυτικής Συμμαχίας η Τουρκία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει γιατί ε, ουσιαστικά έχει εκπνεύσει η διαδικασία η ε, ενταξιακή και θα πρέπει να λήξει και τυπικά και νόμιμα και νομικά, αλλά ας πούμε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία σύνδεσης και να εργαστούμε επικοδομητικά στα πεδία που υπάρχει χώρο συνεργασίας, είτε είναι αυτά οικονομικά, ενεργειακά, τελωνιακή ένωση, ή ε, να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις για την απελευθέρωση θεώσης διαβατηρίων. Είτε είναι αυτό μια κοινή γεωπολιτική συνεργασία, κατά πολέμηση τρομοκρατίας, είτε είναι επιστημονική συνεργασία. Έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα, μια γκάμα θεμάτων, όπου θα μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία και το επιθυμούμε άλλωστε, αλλά έχει δίκιο και η κάτι πύρη. Δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει χωρίς να ε, γίνονται σεβαστές οι αξίες και σε περίπτωση που επαναφέρουν και τη θανατική ποινή, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και συνομιλιών. Η κατάργηση της δημοκρατίας που ισχύει σήμερα αρκεί ε, για να τερματιστούν οι συνομιλίες ενταξιακές. Και θέλω να πω και το εξής. Σκεφτόμαστε και τον Δενίσιο Ξέλ και όλους τους άλλους δημοσιογράφους που ε, έχουν ε, φυλακιστεί. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι και ε, τους κλείνουν φυλακή. Ευχαριστώ. Από την GoNGL, ο κύριος Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Sorry. Uh, for three and a half minutes. Problem, And Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβει κανείς τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία. Νομίζω ότι έχουν λεχθεί πάρα πολύ καθαρά και από την ραπορτέρ, ε, την κυρία Πύρη, και από άλλους συναδέλφους και νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση θα προσθεθούν και άλλες εικόνες. Μόνο δύο λόγια για αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν βαθιά ρήγματα στο τι εστί δημοκρατία στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κρατήσει διάβλους επικοινωνίας ε, γιατί θεωρεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ωφελέσει στο τέλος τον τουρκικό λαό τον τουρκικό λαό που και εμείς ε, νοιαζόμαστε γιατί ε, αυτούς είναι που κυρίως αφορά ε, η δημοκρατία στη χώρα τους. Η σύλληψη και η φυλάκιση εκπροσώπων ενός μεγάλου κόμματος θεωρώ ότι αποτελεί την μεγαλύτερη παραβίαση ε, ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα. Θέλω εδώ να πω ότι ε, εδώ δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Εκπροσωπώ το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Κύπρο που στηρίζει ενεργά και συνειδητά τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού παρά το γεγονός ότι στην κυβέρνηση βρίσκεται ένας άνθρωπος με τον οποίο διαφωνούμε και πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά. Και το κάνουμε γιατί έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι δεν μπορεί η Κύπρος να συνεχίσει διαιρεμένη. Αναφερόμαστε βέβαια σε μια λύση πραγματικής λειτουργικής ομοσπονδίας, τέτοιας που να δίνει όλα τα βασικά δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Εμείς σαν βαθιά παράδοση στη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει κάποια στιγμή θεμελιό στην δημιουργία μιας νέας ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση ε, θα καταλήξει σαν συνολικό κείμενο και τελικό μέσα από πολλές υποθέτω τροπολογίες που θα κατατεθούν και θα κατατεθούν και από εμάς σε όλα τα ζητήματα και βεβαίως σε ό,τι αφορά την ε, Κυπριακή Δημοκρατία και την προσπάθεια επίλυσης. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη φιλοδοξία για τη λύση του Κυπριακού, όμως νομίζω ότι υπολείπεται πολλών βημάτων για να φτάσει η δουλειά της στο επίπεδο της φιλοδοξίας της. Και υπάρχουν τα εργαλεία και θεωρώ ότι ε, πρέπει και μπορεί να αξιοποιηθούν. Έρχομαι στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια υπόθεση που μάλλον από όλους μας θεωρείται ότι είναι σχεδόν χαμένη, εμείς στηρίζουμε την πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας γιατί αυτό θα συνεπαγόταν ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεπάγεται ταυτόχρονα, δεν γίνεται αλλιώς επίλυση του Κυπριακού. Όμως σήμερα το μέγα θέμα είναι η επικαιροποίηση της ε, Τελωνιακής Ένωσης, της συμφωνίας αυτής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που κατά την άποψή μας ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένταξη, εάν θεωρήσει κανείς ότι ε, βρίσκεται ήδη πίσω μας η πιθανότητα ολοκληρωτικής ένταξης, συνολικής ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το θέμα εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να προχωρήσει με παράλληλα ταυτόχρονα θετικά βήματα εκ μέρους της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, τελειώνω με αυτό, εάν επαναλαμβάνω ταυτόχρονα έχουμε θετικά σταθερά βήματα από την Τουρκία προς την κατεύθυνση της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Ευχαριστώ. Thank you. And we go to the green uh, group, Ms. Valero. Ε, Valero. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά τα οποία ακούσανε οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, ιδιαίτερα σε σχέση με την περιγραφή της κατάστασης στην Τουρκία. Η πρόταση η οποία γίνεται από την κυρία Πύρη παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην χώρα αυτή. Δυστυχώς τα πράγματα διαπιστώνουμε πλέον κάθε φορά ότι χειροτερεύουν. Ε, έχουμε φτάσει πια σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την εξέλιξη των σχέσεών μας. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτον, διαπραγματεύσεις για την ένταξη, τελωνιακή σύνδεση και τέλος υπάρχει το θέμα της συμφωνίας εισαγωγικά που έχουμε υπογράψει μαζί τους για το προσφυγικό. Νομίζω ότι ιδιαίτερα με την τελευταία αυτή συμφωνία εμείς ε, προσκυνήσαμε τον κύριο Ερντογάν, ε, τον αγκαλιάσαμε να το πω αλλιώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον βγάλουμε πια από την αγκαλιά μας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η δική μας πολιτική ομάδα δεν έχει καταλήξει σε μια άποψη σχετικά με την διακοπή των διαπραγματεύσεων. Και ένας από τους λόγους είναι ότι τα τελευταία χρόνια εδώ που τα λέμε οι διαπραγματεύσεις δεν είναι και πάρα πολύ δραστήριες, δεν οδηγούν και πουθενά. Έχω την αίσθηση ότι που να πάρουμε μια τελική απόφαση οι διαπραγματεύσεις από μόνες τους θα έχουν σταματήσει. Πάντως, για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ερντογάν αυτό όμως επιθυμεί. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι δεν θα αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση στην παρούσα φάση και τώρα για το προσφυγικό. Θα ήθελα να πω ότι όσο υπάρχει ε, τυπικά τουλάχιστον η συμφωνία αυτή, ο Ερντογάν μας έχει παγιδευμένους. Θα χρησιμοποιήσει και ήδη χρησιμοποιεί τη συμφωνία αυτή κάθε φορά που θέλει να μας εξωθήσει αν θέλετε σε συγκεκριμένες ε, θέσεις και να μας βάλει να κάνουμε αυτά τα οποία δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε θα έλεγα θάρρος και να πούμε ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ε, εμείς δεν θα είμαστε εδώ ε, μόνο και μόνο για να λέμε ότι θα τους ξαναστείλουμε όλους αυτούς στην Τουρκία. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που αναλογεί σε κάθε χώρα. Είναι η μοναδική διαδικασία που θα μας απαλλάξει από την εξάρτηση την οποία έχουμε απέναντι στον Ερντογάν και στο καθεστώς του στην παρούσα φάση λόγω του προσφυγικού. Εμείς δεν θέλουμε επίσης ταυτόχρονα να απομονώσουμε τους δημοκράτες στην Τουρκία που δίνουν μάχη. Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς που δεν θέλουν να συμβούν αυτές οι φρικτές αλλαγές. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το, τα πράγματα στην παρούσα φάση δεν είναι καθόλου εύκολα. Θα υπάρξουν όμως εκλογές το 2019 και δεν ξέρουμε μέχρι τότε πόσο θα έχουν εφαρμοστεί οι αλλαγές αυτές. Πρέπει να στηρίξουμε πριν από οτιδήποτε άλλο τους δημοκράτες. Λοιπόν, ο τελευταίος Κιώδης θα πάρει τώρα το λόγο, αλλά θα πρέπει να κλείσει και ο κατάλογος. Ο κύριος Μποργέτσιο έχει το λόγο για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντίθετα από, τους, από αυτά τα οποία είπε η εκπρόσωπος των Πρασίνων, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα οποία άκουσα από τους προηγούμενους συναδέλφους ε, δεν μου άρεσαν καθόλου, διότι στην ουσία εμείς επιτρέπουμε να χρησιμοποιεί ο Ερντογάν μια ρητορική η οποία ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να τον ακούμε να λέει ότι εμείς διώκουμε τη θρησκευτική ελευθερία, ότι είμαστε ναζιστές, ότι δεν έχουμε σχέση με την δημοκρατία. Ε, όλα αυτά είναι απαράδεκτα γιατί δυστυχώς αυτά αυτός τα κάνει. Συνεπώς λοιπόν ε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε ούτε καν σε σχέση με τη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Να πούμε ότι όταν ελήφθησαν οι αποφάσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να εισακουστούν οι πολιτικές δυνάμεις όπως η ε, δική μου που έλεγαν ότι είναι επικίνδυνο να ξεκινήσουμε μια τέτοια ιστορία ε, με μια χώρα σαν την Τουρκία. Η Τουρκία δυστυχώς σιγά σιγά γίνεται ένα επικίνδυνο Ισλαμικό κράτος το οποίο ε, υποτίθεται ότι μας στέλνει πρόσφυγες αλλά μας στέλνει και κατασκόπους και ταυτόχρονα φυλακίζει ε, τους δημοσιογράφους. Υπάρχει ένας Ιταλός, ε, υπήρχε ένας Ιταλός δημοσιογράφος ο οποίος φυλακίστηκε χωρίς κανένα λόγο και η παρέμβαση διαμαρτυρία της Μογκερίνη ήρθε πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης και να ξεχάσουμε την Τουρκία. Δεν είναι στους μελλοντικού μας προσανατολισμούς. Είμαι ξεκάθαρος. Θα περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο και γι' αυτό ο καθένας θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Ο κύριος Μπρόκ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις ε, στην Τουρκία είναι κάτι που όλοι αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο. Απομακρύνεται η Τουρκία από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προχωρά σε ένα αυταρχικό καθεστώς που δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο του Πούτιν, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Ε, καταπιέζει την ελευθερία της έκφρασης, καταργεί τη διάκριση των εξουσιών και μερικά ακόμα. Και αυτό οδηγεί στο γεγονός να μην πληρούνται ή να πληρούνται και λιγότερο τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Είναι σωστό, πιστεύω, να ακολουθήσουμε τη στρατηγική να μην διαπραγματευόμαστε. De facto έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις και de facto ισχύει αυτό που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πάγωμα. Θα ήθελα όμως να απευθυνθώ στον κύριο Λάμστορφ που μίλησε με μεγάλο πάθος και να πω ότι ήδη από το 2004 ήμουν ε, προς την κατεύθυνση αυτή για τις διαπραγματεύσεις, γιατί τον ξέρω εδώ και καιρό τον κύριο Ερντογάν και ξέρω πού το πάει. Και μου επετέθη το Φιλελεύθερο Κόμμα της Γερμανίας ε, FTP γιατί ε, δεν τα λέω σωστά αυτά για την Τουρκία. Για τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αυτά δεν ορίζουν τις διαπραγματεύσεις, ορίζουν τι πρέπει να πληρεί μια χώρα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δείχνουν επίσης ξεκάθαρα ότι στόχος των διαπραγματεύσεων και παραθέτω περίπου επιλέξει είναι η πλήρης ένταξη ή εάν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή της προενταξιακής διαδικασίας υπάρχουν προβλήματα, ε, ένα διαφορετικό τρόπο διακόπτονται. η εαν κατα τη διαρκεια των διαπραγματευσεων η της προενταξιακης διαδικασιας υπαρχουν προβληματα ενα διαφορετικο τροπο διακοπτονται τερματίζονται. Λοιπόν, εμεί δεν θα πρέπει να ζητούμε να διακοπούν οι διαπραγματεύσει, αλλά ότι αλλάζουμε στόχο και προχωρούμε προ μια κατεύθυνση που δεν ταυτίζεται με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν πληρούνται οι προποθέσει ε, και απαιτήσει που έχουμε εμεί για τη διάκριση των εξουσιών κτλ. Πρέπει να λυθεί και το Κυπριακό. Τώρα έχει την ευκαιρία η Κύπρο που δεν είχε εδώ και πολλά χρόνια να συμφωνήσει, δεν θα πρέπει να ε, απειληθεί και να διακυβευτεί αυτή η διαδικασία και η Τελωνιακή Ένωση επίση ε, θα πρέπει να να Και τελευταία, αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι η Τελωνιακή Ένωση. Γι' αυτό δεν είμαστε έρμεοι στα χέρια του Ερντοάν για τους πρόσφυγες. Και όταν λέμε ότι δεν θα πρέπει να στηρίζουμε τους πρόσφυγες στα 3 εκατομμύρια που είναι εδώ και 4 χρόνια στην Τουρκία, το θεωρώ ε, αν, ανεύθυνες ε, λαϊκιστικές φλιαρίες. Θα πρέπει να στηρίζουμε τους πρόσφυγες στην Τουρκία όπως τους στηρίζουμε και στη ε, Ιορδανία και στο Λίβανο και να μην το καταστρέψουμε. Αυτό νομίζω είναι σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και δημοκράτε, ο κύριο Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη λέχθηκαν πολλά. Συμφωνώ με αυτά που είπε Κάτι Πύρη και μάλιστα συμφωνώ απόλυτα. Οι γραμμές των συζητήσεων περνούν, διέρχονται και μέσω των ομάδων μας. Δεν είναι δηλαδή πάντα σύμφωνες όλες οι ομάδες και εντός των ομάδων. Και αυτό δείχνει ότι οι κατευθύνσει μπορεί να είναι και διαφορετικέ. Πολλά αναφέρθηκαν ήδη και από τον Έλμαν Μπροκ, τα οποία είναι σωστά και σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ μα σχέσει με την Τουρκία. Τώρα, εάν χρειάζεται για να συνεχιστούν αυτά διαπραγματεύσεις, δεν είμαι βέβαιο. Τα θέματα όμως που ανέφερε και ο Λάμστορφ και εσεί, κύριε Μπρόκ, είναι σωστά. Θεωρώ επίση ότι θα πρέπει να συνεχιστούν. Δεν μας απασχολεί η οργάνωση μιας διαρκούς αντιπαλότητας, αλλά η αναζήτηση κοινών τόπων και κοινών συμφερόντων. Άλλωστε είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τους, τους δημοκρατικούς, τους δημοκράτες δηλαδή στην Τουρκία, Επίσης οι δημοκράτες στην Ευρώπη αρχίζουν και μας αμφισβητούν. Πόσο χρειαζόμαστε για να αντιδράσουμε σε πολιτικές απέναντι στην Ουγγαρία για παράδειγμα και μέσα στην, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση στα Βαλκάνια όπου κάποιοι δεν θέλουν πλέον να συμμετάσχουν στις εκλογές, άλλοι δεν δέχονται το αποτέλεσμα των εκλογών οι τρίτοι θεωρούν ότι δεν χρειάζονται πλέον τη δημοκρατία και στα κάνουν όλα μόνοι τους και εμείς και ιδίω το Συμβούλιο των Υπουργών ανησυχεί και ανησυχεί ξανά και ανησυχεί πάρα πολύ και ποτέ δεν ανησυχούσε τόσο όσο σήμερα και ο κόσμος έχει σκάσει τα γέλια με όλη αυτή την υπόθεση. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να σοβαρευτούμε λίγο και να πάρουμε και τους εαυτούς μας σοβαρά υπόψη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ανασταλούν οι συζητήσεις. Με την Τουρκία του Ερντογάν δεν μπορεί να υπάρξει ε, πρόοδος προς την ένταξη. Ευχαριστώ φιλελεύθερη κυρία Σάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απηχώ και εγώ τα όσα λέχθηκαν από την εισηγήτρια σχετικά με τις ανησυχίες, σχετικά με τη διαδικασία του δημοψηφίσματος με συγχωρείτε κάπως, ε, κάποιος με διέκοψε, για τις ανησυχίες του ΟΑΣΕ, της Επιτροπής της Βενετίας, αλλά και την σιωπή της Επιτροπής, όπως είπε ο κ. Φλέκενστάιν και των αρχαίων κατών κυβερνήσεων στη Μάλτα. Εμείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντοτε και σωστά βάλαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά των σχέσεων. Και έχουμε αναφέρει και τις παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών, ω το μέγιστο εμπόδιο για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τώρα, οι προτινόμενες και προβλεπόμενες συνταγματικέ αλλαγέ θα δείξουν ποια θα είναι η πορεία προς το μέλλον. Και εγώ φοβούμαι ότι αυτή η πορεία προς το μέλλον θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην δημοκρατία και στις εμιλιώδεις ελευθερίες των ανθρώπων θεωρώ και εγώ ότι δεν πρόκειται για πολιτική απλά άποψη, αλλά για τις βαρύτατες ανησυχίες οι οποίες προκύπτουν από το δημοψήφισμα. Και θέλω να τονίσω επίσης ότι η εμπιστοσύνη και οι καλές σχέσεις δεν εξυπηρετούνται από δηλώσεις του είδους ότι οι Ευρωπαίοι είναι ναζί και ότι οι Ολλανδοί είναι υπεύθυνοι για μαζική γενοκτονία στην Βοσνία. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδου δημόσιες δηλώσεις τουλάχιστον όχι τώρα. Και το ερώτημα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα. Εγώ φοβούμαι ότι παρόλες τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και του Προέδρου Ερντογάν, διαβλέπουμε να διαγράφεται μία ατζέντα που είναι ρεαλιστική, που βασίζεται στο εμπόριο, στην ασφάλεια, στην φροντίδα των προσφύγων, στην ε, αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όσο σημαντικά και αν είναι αυτά τα θέματα, είναι ωστόσο απαράδεκτο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου, δηλαδή η πραγματική πεμπτουσία των όσων συζητούμε εδώ και έχουμε συζητήσει επί χρόνια, όλα αυτά να κρυφτούν κάτω από το χαλί. Και τα βλέπουμε αυτά και στη βάση των δηλώσεων για τη θανατική ποινή, το monitoring που κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την Τουρκία και ούτω καθεξής. Επιμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλει πρώτο θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ο κ. Παντσέρη για να κάνει ε, την τελική σύνοψη. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες στα πλαίσια των οποίων καλούμεθα να δράσουμε. Κάποιοι ζητούν να είμαστε πιο αυστηροί, κάποιοι άλλοι τονίζουν τα συμφέροντα που έχουμε και τη συμφωνία για τους πρόσφυγες. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση διακοπής, χωρίς να κλείσουμε τις πόρτες, είναι η σωστή γραμμή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε ευφυείς Νομίζω ότι το μοναδικό καθοριστικό στοιχείο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είπε όχι στο δημοψήφισμα και που αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της δημοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παίρνει μέτρα τα οποία θα είναι στο μέλλον αρνητικά για τους δημοκράτες της Τουρκίας Διάβασα άλλωστε τις τελευταίες μέρες ένα σημείωμα του Φερχόφστατ και του Βέμπερ, άλλωστε το είπε, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Λάμπστορφ, ότι θα πρέπει να κλείσουμε την φάση των διαπραγματεύσεων και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι η γραμμή αυτή είναι λανθασμένη στρατηγικά και σε βάθος χρόνου. Αν θέλουμε να έχουμε ένα μήνυμα προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ε, λέγοντας ότι θα σταματήσει η διαδικασία ένταξης επειδή το καθεστώς δεν είναι δημοκρατικό, αλλά θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Αυτό είναι θα έλεγα ένα μήνυμα λανθασμένο ε, και δεν θα πρέπει επαναλαμβάνω να κλείσουμε καμία από τις δυνατότητες που έχουμε ακόμα θεωρητικά μπροστά μας. Ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά ο κύριος Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε πάρα πολύ προσοχή. Την εισηγήτρια είναι πολύ ισόρροπη θα έλεγα, είναι σταθμισμένη η πρόταση την οποία κάνει, χωρίς να αποκρύβει τίποτα. Δυστυχώς ε, υπάρχουν σκιές οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή επικρατούν της ελπίδας. Νομίζω ότι η ανάλυση λέγει ότι έχουμε μια, ένα καθεστώς το οποίο έχει ξεφύγει προς μια κατεύθυνση αυταρχισμού και ως εκ τούτου θεωρώ ότι η κατάληξη της συγκεκριμένης αυτής ε, έκθεσης θα πρέπει να καταλήγει σε κάποιους προσανατολισμούς. Τώρα για τη χειροτέρευση των σχέσεων με την ε, Τουρκία. Αυτό οφείλεται θα έλεγα σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνη η Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι λοιπόν ένα επιπλέον σημείο ισορροπίας, είναι σωστή η επιμονή μας στα κριτήρια της Κοπενχάγης, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση σε επίπεδο προσφυγικό μεταναστευτικό, είναι ευαίσθητο για μας και να δούμε επίσης τι γίνεται και στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με την Τουρκία στα πλαίσια του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Δεν θα πρέπει να αποκρύβουμε όμως τις παραβάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν βέβαια η Τουρκία προχωρήσει στην επανεισαγωγή της θανατικής ποινής είναι σαφές ότι εκεί δεν θα έχουμε κανένα περιθώριο και θα πρέπει να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα. Κατά τα άλλα η έκθεση είναι όπως είπα σωστά σταθμισμένη. Όλα τα στοιχεία της σημερινής κατάστασης λαμβάνονται σωστά υπόψη. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στα αντίστοιχα συμπεράσματα. And Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κ. Παπαδάκης παρακαλώ. Πολύ σωστά η συγγήτρια έχει πει ότι είναι δύσκολες οι σχέσεις με την Τουρκία και θέλω να τη συγχαρώ για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει. Νομίζω όμως ότι ήρθε η στιγμή ως Ευρώπη να δούμε τη σχέση μας με την Τουρκία συνολικά. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ποια ήταν τα λάθη τα οποία διέπραξε η Ευρώπη απέναντι ειδικά στον κύριο Ερτογάν όπου το χαΐδευε για τόσα χρόνια με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αλαζονία του και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας του. Θα είναι καταστροφικό οι σχέσεις της Ευρώπης να εδωθούν μέσα από τις εμπορικές σχέσεις. Και υπάρχουν τέτοιες φωνές. Για να εξυπηρετηθούν οι business. Αυτή είναι η λογική και θα είναι λάθος να αφήσουμε τις όποιες δημοκρατικές δυνάμεις υπάρχουν στην Τουρκία χωρίς να έχουν τη δική μας τη στήριξη και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, να μην εγκαταλείψουμε αυτές τις δυνάμεις, να τις στηρίξουμε. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να δίνουμε στον κύριο Ερτογάν το τυράκι, ούτω ώστε να το πουλά για εσωτερική κατανάλωση στην ίδια τη χώρα του. Το δεύτερο είναι ότι θα κατατεθούν τροπολογίες σε σχέση με το Κυπριακό. Νομίζω Τη στιγμή που η Κύπρος είναι αποκλεισμένη από τον ναυτικό στόλο της Τουρκίας, τον πολεμικό στόλο της Τουρκίας, εκδίδοντας καθημερινά ναύτεξ, οφείλει να καταγραφεί στο ψήφισμα. Και το δεύτερο, πρέπει να υπάρξει θέτε καταδίκη τη τάση τη Τουρκία σε σχέση με τι συνομιλίε. Δεν αρκεί να λέμε μόνο ότι η Τουρκία καλείται να παίξει επικοδομητικό ρόλο. Η Τουρκία ουσιαστικά έχει οδηγήσει τι συνομιλίε σε αδιέξοδο μη αποσύροντας τα στρατεύματα της από την Κύπρο και επιμένοντας να έχει εγγύσεις στη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Then it's για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της και για όλη αυτή τη δουλειά που κάνει με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ με την ε, άποψη που έχει και τη θεώρηση για τη χώρα και τα όσα συνέβησαν το τελευταίο χρόνο. Πολύ σύντομα. Ε, αλλάζει το καθεστώς στην Τουρκία και το κράτος το ίδιο. Δεν είναι μόνο θεσμική η μεταρρύθμιση. Αυτό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα αυτό επιταχύνθηκε και αποκορυφώνεται με την αναθεώρηση του συντάγματος που προφανώς απομακρύνει την Τουρκία από το κράτο δικαίου, την ελευθεροτυπία, τη διάκριση των εξουσιών και τις ευρωπαϊκές αξίες στα πρότυπα και τα κριτήρια της Κοπενχάγη που είναι εκ των όνων κάνευ για την προσχώρηση μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι να κάνουμε. Ακούστηκε ε, διακοπή τη ένταξη γιατί είναι γεγονός ότι ο δρόμος που έχει πάρει η Τουρκία καθιστά ε, αφόρητη, μη βιώσιμη την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πρώτον, ο πολιτικός διάλογος που είχαμε με την Τουρκία ε, ε, ήταν η ε, διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αν φύγουμε από αυτό το τραπέζι, πώς θα συζητήσουμε και πώς θα μπορούμε να επηρεάζουμε τα τουρκικά. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να συνεχιστεί για την ένταξη και θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα. Δεύτερον, τα κονδύλια, τα αναφέρει και η συγκήτρια. Ένας από τους μοχλούς που έχουμε πει στην Τουρκία είναι η προεξιακή βοήθεια. Και το τρία, τρίτο, θα πρέπει να υπάρχει και ένας ελκυστικός ορίζοντας ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην αποθαρρύνεται το μισός πληθυσμός, το 48% που ψήφισε όχι. Και η Τελωνιακή Ένωση είναι ένας τρόπος να δοθεί ε, ένας ορίζοντας. Ο κύριος Λίτς, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι για την πρώτη αυτή έκθεση, το σχέδιο έκθεσή σου. Πραγματικά ε, καλό είναι που συζητούμε σοβαρά ε, τι θα κάνουμε στις μελλοντικές σχέσεις με την Τουρκία. Είπε ο Έλμα Μπρόκο ότι η Τολωνιακή Ένωση είναι το σημαντικό, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα κρίσιμα απέναντι στην Τουρκία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε για την τουρκική διασπορά. Ξέρουμε ότι ε, το Διανέτ που ασχολείται με τα θρησκευτικά θέματα ε, έχει ε, αναγνωριστεί η επιρροή του. Επηρεάζει κάποιους ημάμιδες στη Γερμανία. τώρα έχει σταματήσει αυτή η δράση και τουλάχιστον αυτό είναι αλπιδοφόρο. Ο κύριος Φρόιντ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σαν κάτι για την έκθεση αυτή. Ε, δείχνει πραγματικά ε, μεγάλο θάρρος και το γεγονός ότι βλέπεις μακριά στο μέλλον. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, όχι μόνο γιατί έχουμε απέναντι μας την τουρκική κυβέρνηση, τη οποία τα έργα αποδοκιμάζουμε, αλλά έχουμε και 50% το μισό τουρκικό λαό που είναι από την άλλη μεριά και που περιμένει από μας ε, υποστήριξη. Και εδώ εμείς καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο και είναι ίσως το πιο δύσκολο. Υπάρχει δυνατότητα να διακόψουμε απολύτως ε, τις προεταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά εάν ταυτόχρονα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα βήματα που βοηθούν την τουρκική κυβέρνηση, τότε δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ συζητούμε με μια κυβέρνηση που ταυτόχρονα φυλακίζει εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον ανθρώπους χωρίς την παραμικρή δίκη που ε, καθερεί δικαστές, που ε, συλλαμβάνει και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ό,τι και να έχεις να διαπραγματευτείς με μια τέτοια κυβέρνηση αν το κάνεις δεν είναι και πάρα πολύ ε, σκόπιμη αυτή η δράση ούτε ε, μεγάλη πρόπτικη για το μέλλον. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο φίλος Λάμστορφ και συνάδελφος. Επένεσε τους Αυστριακούς γιατί ήταν οι μόνοι που του είπαν ε, έξω από τα δόντια στη Μάλτα να σταματήσουν διαπραγματεύσεις. Πλην όμως, ε, έχω μια μικρή αντίρρηση εδώ. Δεν πρόκειται για την αυστριακή στάση ε, απέναντι στην Τουρκία, αλλά για λόγους εσωτερικής αυστριακής πολιτικής ακολούθησε αυτή τη στάση. Και αυτό είναι το τραγικό δεν έχουμε στο μυαλό μας την Τουρκία, αλλά τις εκλογές στην Αυστρία που επίκυνται. Αυτά. Καλά εντάξει, και πολλά είπα. Ευχαριστώ. Yeah. Ο Πρόεδρος. Τελευταίος ο μιλητής. Ο κ. Ναβεντές. Ναυρίδης. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η έκθεση εν είναι πολύ διαφοροποιημένη από ό,τι είχαμε δει στο παρελθόν και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, εκτός από κάποια σημεία που θα αναφερθώ. Αλλά σε σχέση με θέματα εκτός Τουρκίας, όπως στη Συρία ή στην Κύπρο, εκεί νομίζω ότι χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για την Τουρκία, δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν διαμορφώνει την τουρκική πολιτική. Την πολιτική της Τουρκίας τη διαμορφώνει ο Ερτογάν. Και οι διαπιστώσεις της Επιτροπής της Βενετίας γύρω από το δημοψήφισμα στην Τουρκία δεν προέκυψαν μετά το δημοψήφισμα, προέκυψαν ένα μήνα πριν το δημοψήφισμα. Και θεωρώ ότι η αξιοπιστία μας θα ήταν σαφώς καλύτερη εάν αναδεικνύαμε την αξία αυτής της έκθεσης πριν από το δημοψήφισμα. Τώρα, για όσα συμβαίνουν εντό Τουρκία, θεωρώ ότι τουλάχιστον μια αναφορά στου κούρδου και άλλου πολιτικού 100, ανάμεσά του 34 γυναίκε που απεργούν, που βρίσκονται σε απεργία πείνα, πρέπει να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε. Τελειώνω όμω με τα εξή. Αναφορές στην Κύπρο. Στο προσχέδιο, και τονίζω, όχι το τελικό κείμενο, το προσχέδιο πέρσι υπήρχε αναφορά και για αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων και για παράδοση της τους του νόμιμους κατοίκους της. Και τα δύο απουσιάζουν. Τελειώνω με την εξή υπόδειξη. The rule of law της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε μια αρχή του ρωμαϊκού δικαίου. Pacta sunt servanda. Οι συμφωνίες στηρούνται. Η Τουρκία λοιπόν έχει δεσμευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη συμφωνία της υφιστάμενης Τελωνιακής Ένωσης με όλα τα κράτη-μέλη και με την Κυπριακή Δημοκρατία και να την αναγνωρίσει. Πώς θα προχωρήσουμε εάν εμείς δεν τηρούμε τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Then we go to the representative of the Commission. Τώρα ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θα ακολουθήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Δράσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο για, το, για τη σημαντική αυτή συζήτηση. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια κυρία Πύρη για το γεγονός ότι το 2016 και η αρχή του φετινού έτους ήταν χρόνια δύσκολα και για την Τουρκία αλλά και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμαστε για την προσπάθεια της ε, ε, εισηγήτριας να καλύψει τα θέματα αυτά με πολύ ισορροπημένο τρόπο. Συμπίπτουν οι απόψει σας με αυτές της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή τη το 2016 για την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από τον περασμένο Νοέμβριο και την ε, δημοσίευση τη εκθέσεώς μας. Συμφωνούμε με πολλές από τις ανησυχίε που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα, στην πρόταση ψήφισματο και τα έχουμε εκφράσει κατά επανάληψη και ιδίω όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, το rule of law, το κράτο δικαίου, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τις θεμελιωδεί ελευθερίες. Όπως είπε και ο Επίτροπος Χάν, εδώ ενώπιόν σας, μετά από την έγκριση των συνταγματικών αλλαγών, έχει έρθει η ώρα για μια ανοιχτή συζήτηση με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το μέλλον των σχέσεών μας. Παρακολουθήσαμε προσεκτικά τα σημεία συγκλήσεως στη συζήτηση της Ολομέλειας την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και πάλι σήμερα το πρωί. Και έχουμε σημειώσει επίσης το γεγονός ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν την κατάσταση στην Τουρκία, στο Γκίμνιχ την Παρασκευή, στο άτυπο ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και θεωρούμε την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στην Μάλτα ναι μεν θετική ως ένα πρώτο βήμα για την ανανέωση του διαλόγου, αλλά ζητούμε τώρα ο διάλογος να επανέλθει στα φυσιολογικά του όρια και να συνεχιστεί γιατί είναι αναγκαίο να, συνε... να ε, γίνεται ο διάλογος σε ισότιμους όρους για το μέλλον της ε, σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με διμερείς συναντήσεις μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και της είπα της εκπροσώπου και του Επιτρόπου Χαν και αναμένουμε να, συνεχιστεί αυτά, να συνεχιστούν αυτά και τις επόμενες εβδομάδες. Η Τουρκία παραμένει από τους πιο σημαντικούς και στενούς μας εταίρους. Οι σχέσεις μας με τη χώρα αυτή εξακολουθούν να είναι πολύ σχηδείς καλύπτουν όλους τους τομείς συνεργασίας. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη συνέχιση της σχέσης αυτής με την Τουρκία, αλλά από σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι ένας γνήσιος, ειλικρινής διάλογος άμεσα με τις τουρκικές αρχές. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, κύριος Πέρες. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήμασταν σιωπηλοί και δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί. Νομίζω ότι τα σχόλια της κυρίας Μοκερίνη μετά τη συνάντηση Γκίμνιχ συμπίπτουν με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην πρότασή σας και ευχαριστώ για την πρόταση αυτή που βρίσκουμε πολύ χρήσιμη. Εμείς ανησυχούμε με τα ευρήματα των ερευνών μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και την κοινωνία γενικότερα στην Τουρκία μέσα από τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και τις πολιτικές μας δηλώσεις. Θέλουμε μια δημοκρατική και σταθερή Τουρκία και μέσω του διαλόγου ελπίζω να το πετύχουμε. Χρειαζόμαστε επαφές eye to eye δεν ξέρω αν το κλίμα στις συναντήσεις θα είναι ευχάριστο ή όχι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση με τους Τούρκους. νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι η Τουρκία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι θέλει να παραμείνει υποψηφία και για να το κάνει αυτό το ξέρει ότι θα πρέπει να σέβεται τα κριτήρια της Κοπενχάγης και σε ό,τι αναφέρεται στο κράτος δικαίου, την δημοκρατία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η εισηγήτρια έχει το λόγο για να κλείσει πλέον την συζήτηση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά όλους τους συναδέλφους. Παρά τις πολιτικές διαφορές τις οποίες έχουμε και παρά τις διαφορές και σε επίπεδο ιδεολογίας Νομίζω ότι μοιραζόμαστε όλοι την ανάλυση της κατάστασης σήμερα. Τώρα να μιλήσω για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι δεν υπάρχουν στην έκθεση. Ξέρετε και γελάει εδώ η, γραμματεία ότι έχουμε κάποιους περιορισμούς με τον αριθμό τον, με το μέγεθος του κειμένου ουσιαστικά. 9.000 γράμματα μπορούμε να βάλουμε. Φυσικά δεν μπορούν τα πάντα να συμπεριληφθούν σε μια τέτοια πρόταση. Κατανοώ ότι ε, και ε, σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με τη Συρία πρέπει να βάλουμε περισσότερα και θα καταθέσω και εγώ τροπολογίες με προθεσμία την 9η Μαΐου. Ε, τώρα, για το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει μια κάποια σαφής διαίρεση. Κάποιοι από εμά δεν ήθελαν ποτέ να υπάρξει μια τέτοια σχέση με την Τουρκία. Άλλοι το υποστηρίζουν αυτό, άλλοι όχι σήμερα. Λοιπόν, ε, πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία σύνδεσης, απλά εγώ υπενθυμίζω την αυστριακή θέση εδώ ε, εγώ αυτό που δεν μου αρέσει η αυστριακή θέση είναι ότι η ίδια η αυστριακή κυβέρνηση, ακόμα και αν η Τουρκία ήταν η πιο δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη, πάλι δεν θα την ήθελε να γίνει μέλος. Ας είστε ειλικρινείς λοιπόν. Είναι καλό το να έχουμε διαφορές, αλλά είναι κακό το να κρυβόμαστε πίσω από το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Είτε μας αρέσει είτε όχι η διαδικασία αυτή, συνθήκη τι λέει, λέει ότι αν υπάρχει μία συστηματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, στην κάθε χώρα θα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η συνθήκη τι λέει, λέγει ότι αν υπάρχει μια συστηματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, στην κάθε χώρα, θα πρέπει να υπάρξει διακοπή των διαπραγματεύσεων και υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντί να μιλάμε θεωρητικά λοιπόν ε, για το ποια θα είναι η μελλοντική μορφή των σχέσεών μας θα πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε μια ενότητα θέσεων στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Τώρα για τις πιστώσεις. Όπως βλέπετε και στην πρόταση ε, είπα ότι όσαν υπάρξει μια διακοπή των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρξει και διακοπή των ε, πιστώσεων, της ροής πιστώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί μαζί με την Άγκυρα και αν κάποιοι από εμά θέλουν να υποστηρίξουν τους δημοκράτες στην Τουρκία, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για επίσημη διακοπή θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε με τις πιστώσεις αυτές. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις για να βοηθήσουμε τους δημοκράτες και τον πληθυσμό στην Τουρκία. Ε, Μία συνάδελφος είπε ότι εμείς εδώ δεν συζητάμε για ένα πολιτικό όραμα ε, η διακοπή των διαπραγματεύσεων. Είναι μια απλή συνέπεια του τι συμβαίνει με την Τουρκία και στην Τουρκία πολλοί Τούρκοι λένε ότι δεν σέβεστε το αποτέλεσμα των, του δημοψηφίσματος. Το θέμα δεν είναι η διακοπή, ε, το ότι δεν πιστεύουμε εμείς το δημοψήφισμα και ε, απλά εξηγούμε ότι έχει συνέπειες το δημοψήφισμα αυτό ε, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για το Κυπριακό, όπως γνωρίζετε, <coughs> γνωρίζουν οι συναδέλφοι, είχα πάει στη Λευκοσία όταν είχαν διακοπεί προσωρινά οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Χαίρομαι που ξεκινούν πάλι, κατανοώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία και απαιτείται η πλήρης στήριξη από πλευράς όλων και φυσικά και από πλευράς Τουρκίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτή η, αυτό το πρόβλημα τόσες δεκαετίες να α, καταλήξει κάπου προς όφελος όλων των κοινοτήτων. Πέραν αυτών έχουμε αρκετά κοινά στις προτάσεις που άκουσα, αλλά αν εμείς πιστεύουμε ότι η Τελωνιακή Ένωση είναι ο μοχλός, εσείς οι πράσινοι γιατί δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο μοχλός αυτός. Πώς θα βοηθήσουμε τους δημοκράτες στην Τουρκία αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και εδώ εννοώ την Τελωνιακή Ένωση. Πώς θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω. Μια μικρή αντίδραση σε αυτά τα οποία άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εκτιμώ αυτά τα οποία έχουν κάνει, αλλά σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι το μήνυμα που στείλαμε στον Επίτροπο Χάν πέρυσι είναι no business as usual και νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει κάθε φορά να περιμένει ξεκάθαρα το τι θα κάνει κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να συντάξει μια αξιολόγηση του πώς έχει η κατάσταση σε επίπεδο κριτηρίων της Κοπενχάγης. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει κάποια μέτρα το ταχύτερο δυνατόν για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, εάν τώρα δούμε τις ανακοινώσεις ε, της υπηρεσίας αυτής βλέπουμε ότι υπάρχει υλικό για να μας κάνει να ανησυχήσουμε. Το μήνυμα το οποίο απεστάλλει από τη Μάλτα έγινε αντιληπτό στην Τουρκία σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίζει τα λάθη της. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ε, τότε δεν ήταν ένα σωστό μήνυμα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Μάλτα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μπήκαν στον κόπο να κάνουν τις προτάσεις αυτές και θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις με τους Σκιώδης και ελπίζω σαν κοινοβούλιο να καταλήξουμε ε, σε μια ε, καλή πρόταση. Και τέλος, για να διευκολύνουμε την εξέβρεση συμβαστικών προτάσεων θα βοηθούσε πάρα πολύ αν Κάνετε τις τροπολογίες σας στα αγγλικά οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ξέρω ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να τις γράφετε στη γλώσσα σας, αλλά θα βοηθήσει τη διαδικασία πάρα πολύ αν φέρετε τις τροπολογίες στα αγγλικά για να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι βέβαιος ότι έχετε πολλή δουλειά ακόμη. Για να σας διευκολύνω θα επαναλάβω ότι... Α, με συγχωρείτε εσείς κύριε Λάμστορφ. Πολύ σύντομα διότι έγινε παρατήρηση προσωπικά για εμένα και ο κανονισμός μου επιτρέπει να απαντήσω. Ο Έλμαρ Μπροκ λάθος κατάλαβε. Εγώ δεν μιλούσα για τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αλλά για το negotiating framework, για το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Περί, αυτό, περί αυτού πρόκειται. Έλμαρ, έχεις δίκιο, και θα πρέπει να προσέξεις καλύτερα τι λέω, έχει δίκιο. Ήδη όμω ο μέγα φιλελεύθερο Κόνραντ Άντεναουερ είχε πει ότι και ο πολιτικό αντίπαλο δεν μπορεί να μα. Ε, αποτρέψει από το να γίνουμε σοφότεροι μέρα με την ημέρα. Έχεις δίκιο λοιπόν μεν, ε, αλλά η θέση μας έχει αλλάξει. Ευχαριστώ. Σύντομη παρατήρηση μιας και ακούστηκε το όνομα του κυρίου ε, Μπροκ. Πάντα μας ξεπερνούν ο Λάμστοφ και η Φιλελεύθερη. Δηλαδή προσαρμόζονται ταχύτερα στην κάθε κατάσταση. Καλά, ελπίζω ότι διευκρινίστηκαν ε, τα προσωπικά. Θα επαναλάβω ότι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 9 Πέμπτου, 9 Μαΐου, 6 το απόγευμα και ελπίζω να επιτύχετε να περάσουν και οι συμβαστικές σας τροπολογίες καθώς θα προχωρούμε. Κλείνουμε το υπαριθμό 4 λοιπόν και ερχόμαστε στο υπαριθμό 5, σύσταση προς το Συμβούλιο, συστάση προς το Συμβούλιο για την 72η Σύνοδο Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σας υπενθυμίζω σε όλους ότι κάθε χρόνο η ΑΦΕΤ συντάσσει συστάσεις του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να διοχετευθούν στις προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 72η εν προκειμένου Σύνοδο Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Τι συστάσει αυτέ και τι προτεραιότητε θα τι εγκρίνει το ε, Συμβούλιο τον Ιούλιο. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έχουμε λάβει 225 τροπολογίες. Η συνάντηση των σκιωδών θα γίνει αύριο για να συζητηθούν συμβαστικέ τροπολογίες οι οποίες έχουν ήδη διανεμηθεί από την Γραμματεία. Είναι παρόν ο κύριος Μαρινέσκου, ο οποίος ε, θα τοποθετηθεί αντικαθιστώντας τον κύριο Κόβατσεφ που είναι ο εισηγητής. Θα συζητήσουμε και τις τροπολογίες. Το δε σχέδιο θα συζητηθεί αύριο στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνει σε μια αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κ. Μαρινέσκου για να μπορέσει να ε, αναπτύξει τις απόψεις του εισηγητού κ. Κόβασεφ. Δεν είναι παρόν, λέει η κυρία Μανέσκου, εγώ είμαι η κυρία Μανέσκου, ο κύριο Μαρινέσκου είναι αλλού, δεν είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών. Βέβαια τα ονόματά μας ε, μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε σύγχυση. Ο συνάδελφός μου Κόβατσεφ, που είναι εισηγητή, δεν μπόρεσε ε, να προσέλθει σήμερα διότι είχε κάποιες επίγουσες ε, υποχρεώσεις. Θα διαβάσω λοιπόν την δήλωσή του. Θα ήθελε πρώτα να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες τα μέλη τη ομάδα εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Εθνών, σκιώδη ηγητέ πολιτικού συμβούλου για την επικοδομητική του προσέγγιση, καθώ επίση και την γραμματεία τη Επιτροπή ΑΦΕΤ. Υπενθυμίζει ότι πέρσι επανήλθαμε στην παραδοσιακή μορφή ετησίων συστάσεων προ το Συμβούλιο, με στόχο να διοχετευτούν τα, τα σχόλια αυτά στην προετοιμασία των ε, προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν συστάσεις προς το Συμβούλιο για ειρήνη ασφάλεια, για τον αφοπλισμό, για την μετανάστευση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ανάπτυξη, τις αλλαγές του κλίματος και την αναθεώρηση του συστήματος των ΗΠΑ. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 225 τροπολογίες. Μέχρι τώρα δεν έχουμε φέτος έκθεση της Επιτροπής, Περιβάλλον, της Επιτροπής Αναπτύξεως μάλλον, Έχουμε όμως κάποιους γενικούς στόχους. Επίσης υπάρχουν πολλές τροπολογίες με παρόμοιο περιεχόμενο, τις οποίες θα περιλάβουμε σε συμβαστικές. Θα γίνει συνάντηση το σχεδόν αύριο και ελπίζει ο εισηγητής ότι θα είναι επικοδομητική η προσέγγιση τους όπως πέρσι όπου τέλειξαν τελικώς σε 22 μόνο συμβαστικές τροπολογίες. Αύριο θα συναντηθεί επίσης η ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Ορισμένες από τις τροπολογίες αναφέρονται σε, στην διασφάλιση ότι η Γενική Συνέλευση σε συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ θα δώσει όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε μια λύση στην βάση των δύο κρατών ε, μέσα στα πλαίσια των ε, συνόρων του 1967 με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών, με ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ούτω καθεξής. Επίσης, η responsibility to protect να παραμείνει βασική αρχή των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη και ούτω Να ενισχυθούν δράσεις για την ε, αύξηση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στην εξτρεμιστική προπαγάνδα για οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά θέματα, να ζητήσει από τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών να συμμετάσχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, κυρώνοντας το καταστατικό της ε, Ρώμης καθώς και της τροπολογίας της Καμπάλα, να λάβει ε, έδρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας, να αποφύγουν να χρησιμοποιούν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας το δικαίωμα βέτο που διαθέτουν σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, να ενισχυθεί ο Γενικός Γραμματεύς των ΗΠΑ στην τροποποίηση, στη μεταρρύθμιση που επιφέρει στην αρχιτεκτονική των ΗΠΑ, να απλουστευτεί η λειτουργία της γραμματείας με αποκέντρωση και ευελιξία και να δοθεί μια καλύτερη, απλούστερη μορφή στις ε, στην οργάνωση του, ε, των οικονομικών του Διεθνούς Οργανισμού. Αυτά θα γίνουν το Σεπτέμβριο, τότε θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Επειδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί η άποψη της ε, ΑΦΕΤ μέχρι τα τέλη του Μαΐου, για να μπορέσει να δοθεί η σύσταση τον Ιούλιο. Εισηγητή ελπίζει ότι θα βρείτε την έκθεση και τι συμβαστικέ τροπολογίε στι οποίε θα καταλήξουν αύριο και οι Συγητές επικοδομητικά και ότι θα μπορέσετε να την υποστηρίξετε στην σχεδιαζόμενη, στην ε, προβλεπόμενη μάλλον, ψηφοφορία τη ΑΦΕΤ στι 30 Μαου. Ζητώ συγγνώμη για το λάθο μου με το όνομά σα, λέει ο πρόεδρο. Τώρα, σοσιαλιστέ και δημοκράτε, ο κύριο Φρόιντ, ο οποίο επίση αντικαθιστά τον αρμόδιο σκύρι Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που αντικαθιστώ την κυρία Πόστη για μια έκθεση που είχα ζητήσει εγώ να αναλάβω στην αρχή. Εν πάση περιπτώσει, ευχαρίστω θα διαβάσω αυτά που λέει. Και πρώτα, η Σοάια Πόστ ζητεί συγγνώμη που είναι απούσα σήμερα λόγω άλλων υποχρεώσεων. Ευχαριστώ την εισηγήτρια εξ ονόματός της εν προκειμένου, εν προκειμένου βέβαια τον εισηγητή και ο Κόβατσεφ για την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση του. Έχω ορισμένα σχόλια για τις τροπολογίες της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών για την ειρήνη και ασφάλεια, τον ρόλο των γυναικών και με πολλές τροπολογίες έχουμε ε, προσπαθήσει να τονίσουμε ε, τον ρόλο των γυναικών όλα αυτά μέσα στα πλαίσια και των ψηφισμάτων της, των ΗΕ με δραστηριότητε οι οποίες θα αποκαθιστούν την ισότητα μεταξύ ανθρώπων και γυναικών. Έχουμε επίσης ορισμένες τροπολογίε για την χρήση της αρχής responsibility to protect. Για θέματα όπως προσφυγικό, μεταναστευτικό, πρόσφυγες λόγω κλιματικών συνθήκων κλπ. χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα θέματα αυτά και να υπάρξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Ζητούμε να υπάρξει η ειδική συζήτηση για τους πρόσφυγες για λόγους αλλαγής κλίματος και επειδή αυτό θα γίνει όλο και εντονότερο το θέμα λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας θερμοκρασίας χρειάζεται λοιπόν να ληφθεί μέρημνα. Αγώνας κατά της θερμοκρατίας Οι τροπολογίες της ομάδας S&D τονίζουν τη σημασία της συμπερίληψης του κράτους δικαίου στις ε, αντιτρομοκρατικές δράσεις που θα πρέπει να αποτελεί και το βασικό πυλώνα των δράσεων αυτών. Για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία χρειάζεται ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ε, τοπικών κοινοτήτων για τον αφοπλισμό και την μη διάδοση των εξοπλισμών. Θέλουμε να υπάρξει νομικό πλαίσιο στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου για μη επιδρομένα αεροσκάφη καθώς και ε, οπλισμένα ρομπότ. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για το θέμα αυτό και για το προσεχές μέλλον. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου. Οι τροπολογίες μας τονίζουν κατ' επανάληψη την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων και ιδίω παιδιών, νέων και γυναικών και να τους δοθεί η δυνατότητα να παίξουν το ρόλο των φορέων της αλλαγής σε ένα πλαίσιο αποκατάστασης της ειρήνης. Σε ό,τι αφορά πρόσωπα LGBT. Χρειάζεται ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και προστασία των ομάδων αυτών. Με ενθάρρυνση της, ε, των δράσεων κατά οποιασδήποτε προσβολής τους. Το κείμενο αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα ηθαγενών πληθυσμών και πληθυσμών Ρωμά και ζητεί από τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμόσουν τις συστάσεις του ειδικού εισηγητού των ε, Ηνωμένων Εθνών για θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, ε, ρατσιστικών διακρίσεων και δυσανεξίας. Να κάνω και ένα διάλειμμα για να προλάβουν να πάρουν αναπνοή οι διερμηνείς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τα ε, αναπαραγωγικά δικαιώματα με διεθνικές πρωτοβουλίες και για πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου για δράσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ASCBD. E Τώρα, κάπως είναι μακρύ το κείμενο, ε, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Στήριξη του, είπα, του αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση ε, των ε, καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδίως σε περιπτώσεις σημαντικών παραβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα των επιχειρήσεων. Υποστηρίζουμε επίσης ένα διεθνώς δεσμευτικό νομικό όπλο στάσιο για το μέλλον. Και τέλος, για την ε, αναμόρφωση του συστήματος των ΗΠΑ. Η ομάδα μας ζητεί να τροποποιηθεί ο οργανισμός των ΗΠΑ για να αντιμετωπίζει καλύτερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η τροπολογία του Γιολάινεν ζητεί να υπάρξουν κοινέ θέσεις στο UNSC. Ο στόχος μας πάντως είναι να υπάρξει μία ενιαία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ζητήσουμε αναμόρφωση του, του, της χρήσης του δικαιώματος βέτο όταν υπάρχουν ε, παραβιάσεις των ε, ε ανθρώπινων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. τέλος, όλοι αναμένουμε την στενή συνεργασία με τον εισηγητή και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες στην επερχόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ο κ. Κίσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριο Σκιουτσούκ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή κύριο Κοβάτσεφ για τις προσπάθειές του ε, για ε, τη σύσταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει ένα κατάλογο κοινών προτεραιοτήτων εν ώψη της ε, επικείμενης ε, Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 255 τροπολογίες με στόχο να αυξήσουν την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν συμφωνούμε για τα παγκόσμια ζητήματα πάντα, και σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μία φωνή και να συνεννοηθούμε ε, στα θέματα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πιο αφοσιωμένους ε, ε, υπερασπιστές και αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτισμικές ελευθερίες, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των λαών. Ωστόσο θα πρέπει να εξακολουθεί να υποστηρίζει αυτές τις πολυμερείς προσπάθειες για να έχουμε λύσεις ε, και βιώσιμη λύση του συνεχιζόμενου προβλήματος στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, τα διεθνή ε, σύνορα και την εδαφική ακαιρεότητα των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτιού Καυκάσου. Ε, και να ε, βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση συνεχιζομένων ε, σειράξεων. Τέλος, θα πρέπει να διατρανώσουμε την πάγια και διαρκή υποστήριξή μας στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, όχι μόνο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με άλλες δράσεις που διαφυλάσσουν την φύση, την προστατεύουν και βελτιώνουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς, εξ ονόματος της Νοτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης αυτής και ομολογώ ότι πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους με βρίσκουν σύμφωνο. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή όλων μας στη συζήτηση αυτή ότι δύο είναι οι βασικές προκλήσεις μάλλον. Αν δούμε την ε, συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με το Brexit, με τις αυξανόμενες ε, ε, θέσεις των κρατών μελών που υπερασπίζονται εθνικά ζητήματα και συμφέροντα, θα πρέπει να συζητήσουμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να έχει και μεγαλύτερες δυνατότητες και ικανότητες δράσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, να υποστηρίζει προσεγγίσεις προς την επίλυση ε, συγκρούσεων. Δηλαδή, να κοιτάξουμε το κεφάλαιο αυτό που αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συνολικότερο θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να έχουμε μία έδρα ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας μόνιμου μέλους και πώς θα την επιτύχουμε αυτή. Συμφωνώ με τον Γιολάεν και την ε, ε, Μπάρμπαρα Λόχμπίλερ στην τροπολογία τους, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη διεκδίκηση και πώς θα τη δούμε στο επόμενο 18 μήνο. Ο περιορισμός του δικαιώματος ε, βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να είναι μια τέτοια δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να το συνδέσουμε και με το γεγονός ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πρέπει να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή για την επίλυση των συγκρούσεων και των σύραξεων. Ως ομάδα εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες αυτές, να τις συζητήσουμε. παρόλα αυτά θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε και στην καθημερινή μας κοινοβουλευτική δουλειά και σε άλλα θέματα και σε άλλες εκθέσεις για να καταλάβουμε ότι αυτό υποστηρίζει την προσπάθεια που καταβάλουμε στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα ήθελα να θέσω υπόψη είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, να ενισχύσουμε εκείνα τα κεφάλαια στην έκθεση που αναφέρονται στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη, στην κλιματική αλλαγή κλπ. Διότι αν δείτε τις λεπτομέρειες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη διεθνή πολιτική και στις διεθνείς μας σχέσεις, στη μεγάλη τους πλειονότητα πηγάζουν από αυτή την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν κάνει κάποιες τροπολογίες για την έκθεση αυτή, ε, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Προσβλέπω λοιπόν στην πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία στην ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις θετικές εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν και να εμπλουτίσουμε πολύ όλη την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάδα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχει ένα συγκρότημα από τη Σκοτία γνωστό ροκ που λέγεται Ντελαμίτρη και το τραγούδι τους λέγεται Nothing ever happens, δεν τρέχει ποτέ τίποτα. Λοιπόν έτσι φαίνεται και εδώ και νομίζω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε και με την αρχική έκθεση του κύριου Βαρίνεν και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει τακτική και να προχωρήσει για την υπόθεση αυτή στο Σύμβουλιο Ασφαλείας. Η δική μου χώρα αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε και τον κύριο Σόλτς Πολλές φορές η δική μου ομάδα συμβαδίζει με τη δική σας κύριε Σόλτς και αυτό είναι περίεργο, αλλά είπατε ότι υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης των εθνικισμών και εγώ θα προσέθετα και το λαϊκισμό. Νομίζω ότι εγώ είμαι υπέρ της αποχώρησης της χώρας μου από την Ένωση γιατί ακριβώς έβλεπα καθώς βυθιζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίσεις την άνοδο των εθνικισμών. Υπάρχουν πολλά διακυβεύματα στις διάφορες χώρες, στις 27 χώρες και κάποια στιγμή θα έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό είναι σημαντικό το θέμα και συμβαίνει μάλιστα και στα πλαίσια μιας εκλογικής εκστρατείας στη Γαλλία που δίνει την ευκαιρία και στην κυρία Λεπένα να διεκδικήσει την Προεδρία. Θα πρέπει λοιπόν η αντίδραση από εδώ και πέρα να έρθει από τη Γαλλία γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει οπότε θα κρατήσει τη θέση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας να δούμε ακριβώς τι γίνεται με χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικές μεταξύ τους για τον τρόπο με τον οποίο θα δράσουν οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε το βάρος μας στα Ηνωμένα Έθνη και να πιέσουμε ακριβώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση ε, μια χώρα σαν την Σουηδία να γίνει η θέση της σεβαστή και να εκφραστεί σαν κεντρική θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς λοιπόν εγώ θα καταψηφίσω την συγκεκριμένη έκθεση. Ε, ε, ε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν κατέθεσα τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Έχασα την ευκαιρία. Ε, θα ήθελα όμως να λάβουν υπόψη οι σκιώδεις και ο εισηγητής κάτι σημαντικό στην αυριανή του συνεδρίαση. Και βέβαια με τις τροπολογίες ε, θα ε, αναφερθεί περισσότερο η υπόθεση της ανάπτυξης και θα αναπτυχθεί περισσότερο φυσικά. Απλώς να δούμε τι κάνει το Κοινοβούλιο και πώς εργάζεται στα πλαίσια ε, των φορολογικών ζητημάτων ε, και ε, των δύο εξεταστικών επιτροπών που είχαμε για τα και για τα Panama Papers, τα έγγραφα του Παναμά. Εκεί ακούσαμε εμπειρογνώμονες από τις αναπτυσσόμενες χώρες και μας είπαν ότι η καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίων είναι απολύτως κρίσιμη και αποφασιστική έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια. Και επίσης αυτό συνδέεται ξεκάθαρα και με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλήματος βραμικού χρήματος, της τρομοκρατίας και προφανώς όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πρέπει να εθαρρύνουμε όσο και να υποστηρίξουμε τις υφιστάμενες προτάσεις να συσταθεί ομάδα εργασία σε επίπεδο ΟΗΕ που να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έγιναν προτάσεις το 2015 στη Σύνοδο Κορυφής για την Ανάπτυξη του ΟΗΕ, αλλά μετά, κατά μυστήριο τρόπο, όχι και τόσο μυστήριο μάλλον, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαν και τον μποϊκόταραν αυτό. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δείξει λοιπόν ηγετική στάση ε, και πράττοντας ε, κάτι τέτοιο θα την... Ε, δηλαδή ένα κεφάλαιο για, το περιβάλλον, για το, την ανάπτυξη. Ο κύριος Μπέρανεν από την Σπρασένους, Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιρενεν. Καλή έκθεση του κύριου Κοβάτσεφ για συζήτηση σε αυτό το σχέδιο έκθεσης δίνεται μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και πάλι. Και από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η τάση που επικρατεί τώρα στην Επιτροπή μας και σε όλο το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ μικρή η προσοχή που αφιερώνεται σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει κάθε είδους πολυμερή παγκόσμια συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγετική δύναμη στην προσπάθεια αυτή σε τομεί όπως είναι εμπορική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, περιβάλλον. Και αυτά τα ζητήματα κατά την άποψή μου θα πρέπει να αναφέρονται περισσότερο σε εκθέσεις μας για τα Ηνωμένα Έθνη και ε, τη Γενική Συνέλευση. Εγώ έχω υποβάλει αρκετέ τροπολογίες για να ενισχυθεί ε, η αναπτυξιακή πολιτική και η μεταρρύθμιση του συστήματος των ΗΕ, να αφαιρθεί ο ρόλος της, ε, του ΕΚΟΣΟΚ του Συμβουλίου ε, Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων που να έχει μια ισχυρή παρουσία για τα αναπτυξιακά εκτός από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει όμως να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον σε τέτοιου είδους εκθέσεις, σε όλους τους άλλους τομείς Εντάξει, είναι σημαντική η ασφάλεια, αλλά υπάρχουν και τα άλλα σημεία. Και η παγκόσμια συνεργασία έχει επιπτώσεις στην πολιτική ασφαλείας. Προσβλέπω λοιπόν στις εργασίες της ομάδας της για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών και εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων του συστήματος των Εθνών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι για την αυριανή συζήτηση έχει σημασία το εξής. Ε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, θα πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερο χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα δεν έχουμε στρατηγική, άρα υπάρχουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και πέρα από τις εκκλήσεις που κάνουμε να αυξηθεί η, η προβολή και των διαφόρων πολιτικών που θα πρέπει να διέπονται από αυτούς τους στόχους. Αυτό θα το πούμε και στον συνάδελφο που εκπονεί την έκθεση για τον προπολογισμό που είναι το επόμενο δημοσιονομικό έτος. Ωραία. Τελειώνει το κατάλογο των ομιλητών. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, μέχρι αύριο συνεχίζεται η συνεδρίαση των σκιωδών των 20 του μηνός ψηφίζουμε και τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Έχουμε το 6 που είναι το επόμενο θέμα μας και το έχουμε προβλέψει για τις 11, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ δεκάλεπτο. λεπτό, ραντεβού στις 11 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 yes, I think the clock is approaching 11 o'clock, so we will... Επειδή η ώρα πάει 11, νομίζω καλά θα κάνουμε να επαναλάβουμε τη συνεδρίαση. Έχει έρθει και ο εισηγητής, όλα καλά. Είμαστε στο σημείο 6 λοιπόν. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής τη σταθερότητα και την ειρήνη. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας μετά τη συζήτηση με την Υπηρεσία Εξωτερικής δράση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 21η Μαρτίου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή. Sí, Κύριε Σντάνζο. Δεν θα μακρηγορήσω. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα αυτό δεν υπάρχουν ε, πολλές ε, τροπολογίες και για λόγους μορφής και για λόγους ουσίας. Καταρχάς το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και δεν υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις. Επί της ουσίας πρέπει να πω ότι ε, το πρόβλημα είναι αρκετά επίγον. Έχουμε καθυστερήσει. Καλούμεθα να εκφραστούμε πάνω σε ένα μέσο το οποίο το Συμβούλιο θα ήθελε να θέσει σε εφαρμογή ήδη εδώ και πολλά χρόνια οι δράσεις και οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περιμένουν αυτό επίσης εδώ και πολλά χρόνια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία δεν εξαρτάται, δεν εξαρτώνται από μας και το δείχνουν αυτό οι τροπολογίες που έχουμε. Υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή λοιπόν με τους σκιώδεις απόψεων Ήδη έχω λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει επί των τροπολογιών που έχω ήδη προτείνει και γι' αυτό στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τους σκιώδεις θα ξανακάνω κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν από την ομάδα των Πρασίνων, των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελευθέρων. Νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεων την οποία είχαμε μέχρι τώρα μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκληση των αναλύσεών μας. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι εμείς δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή μία πρόταση εκθέσεως, αλλά μία τροπολόγηση κανονισμού, δηλαδή νομικά και πολιτικά είμαστε σε ένα πάρα πολύ ε, δεσμευτικό πλαίσιο. Φυσικά και υπάρχει διάθεση και την κατανοώ να γράψουμε εκ νέου αν θέλετε, να σχεδιάσουμε εκ νέου την σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι επί του παρόντος η δουλειά μας. Εμείς θέλουμε να καταστήσουμε τον κανονισμό αυτό όσο περισσότερο γίνεται λειτουργικό και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ δεν θέλησα να γράψω εκ νέου, αν θέλετε, την πρόταση αυτή. Μετά λοιπόν από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων την οποία είχαμε, ελπίζω να καταστεί δυνατό να μπορέσουμε ε, να μέσω λίγων τροπολογιών να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Σκιώδης τώρα. Σοσιαλιστές και δημοκράτες δεν βλέπω ε, τον σκιώδη εισηγητή, οπότε θα δώσω τον λόγο στον εαυτό μου. Με μεγάλη γενναιοδόρια για το χρόνο αγόρευσης. Θα είμαι σύντομος όμως όλα αυτά. Ήδη συνεδρίασαν οι σκιώδεις εισηγητές. Η ομάδα μας συμφωνεί με τον εισηγητή η έκθεση δεν θα πρέπει να ε, είναι πάρα πολύ περιοριστική, είναι πρακτική σημασία. Πρέπει η έκθεσή μας να είναι ένα εργαλείο που να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όχι καμιά φιλοσοφική τοποθέτηση και δοκίμιο που να είναι πολύ ωραία αλλά να μην μπορεί να εφαρμοστεί στον πραγματικό κόσμο. Θα συνεννοηθούμε και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Είμαστε πάντως σε κοινή γραμμή με τον εισηγητή και στόχος είναι να κινηθούμε γρήγορα και με ευελιξία. Σταματώ εδώ και δίνω το καλό παράδειγμα και πάμε στον επόμενο σκιώδη εισηγητή. Και τώρα κατέφθασε ο συνάδελφος σοσιαλιστής και δημοκράτης ο εισηγητής, ο κύριος Μαμίκινς. Uh, um, ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση αυτή βοηθάει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το δικό της προϋπολογισμό την αντίστοιχη δράση. Είναι επαναστατική πρόταση. Μπορούμε να επιτύχουμε στόχους ε, ασφάλειας ε, σε ε, τρίτες χώρες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά χρειάζεται προσαρμογή για να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε μία από τις βασικές αρχές της, του ανθρωπιστικού δικαίου Δηλαδή βοήθεια να, μην, είναι βοήθεια και να μην είναι επιζήμια. Ε, επίσης, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε κάθε φορά αν υπάρχει ένα πρόβλημα ασφαλείας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα και αν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακή βοήθεια χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ασφαλείας πρώτα. Η δεύτερη ερώτηση, έχουμε πολιτική στήριξη. Εκείνοι που στρέφονται κατά της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Πώς δηλαδή θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ασφάλεια των αναπτυσσομένων χωρών χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς προβλήματα από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού. Και αν δεν έχουμε βιώσιμε εναλλεκτικέ προτάσεις, να συζητούμε τα κριτήρια τη συγκεκριμένη πρόταση και τι προϋποθέσεις. Ας πούμε, ποιε είναι οι συνθήκες που επικρατούν. Έχουμε τις οδηγίες του ΑΣΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια δηλαδή. Και έχουμε και την ατζέντα το 2030 του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στόχους ασφάλειας, ε, ειρήνης και δικαιοσύνης. Άρα πρέπει να ενισχύονται οι θεσμοί σε ευαίσθητες έφθραυσες χώρες, χώρες που πλήττονται από σειράξεις. Ε, τι ε, πραγματογνωμοσύνη χρειάζεται, ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο του μηχανισμού και τη διαδικασία. Για να υπάρξει λοιπόν αυτό ο μηχανισμό να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να βρούμε απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση και σε άλλε. Εμεί είμαστε στη διάθεσή σα να συζητήσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Οστρεβίσιους θέλει να πάρει το λόγο ξέρω με του σκιώδη εισηγητή τη ομάδα των φιλελευθέρων. Μάλιστα, έχω το προνόμιο να μιλώ εξ ονόματος της συναδέλφου Χίλντε Βάουτμανς που δεν μπόρεσε να φτάσει εγκαίρως στην Επιτροπή μας σήμερα το πρωί και μου έστειλε το κείμενό της να το διαβάσω. Ως φιλελεύθεροι χαιρόμαστε για το μηχανισμό συμβολής της σταθερότητα και την ειρήνη και την αναθεώρησή του για να δούμε ε, ποια θα είναι η δράση των στρατιωτικών φορών που πρέπει να είναι περιορισμένη ε, σε έκτακτες περιστάσεις. Συμφωνούμε με τον εισηγητή κύριο Ντανζάν ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό και απαραίτητο. Επίσης ε, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους υποστήριξη μπαίνει πλέον στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε την πρόθεση να καταθέσουμε τροπολογίες που θα επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στο σχέδιο έκθεση του κυρίου Ντόνζα. Ωστόσο, θα υποβάλουμε τροπολογίες για να διευκρινιστεί και να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογή της πρότασης, Ποιε θα είναι ασφαλιστικέ δικλείδες, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης ε, στρατιωτικών ε, παραγόντων με ασφαλιστικές δικλείδες χέγγια και κατευθυντήριες γραμμές. Ωραία. Προχωρούμε. GoNGL, ε, η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Με ταχύτητα και με ευκαμψία αυτή είναι η περιγραφή της συζητήσεως που κάνουμε εδώ τώρα. Ο εισηγητής, ο κύριος Ντανζόν, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις εκφράσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας δείξει ότι πρόκειται μια καθαρά τεχνική συζήτηση. Ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το ταχύτερο δυνατό να μπορέσει το εργαλείο αυτό να καταστεί, να να καταστεί ε, χρησιμοποιήσιμο. Άκουσα από να μιλούν για επαναστατική απόφαση. Ας το ξανασκεφτούμε λιγάκι αυτό, έστω και αν η μεν και η δε εννοούμε διαφορετικά τις επαναστατικές εξελίξεις. Πρόκειται όντω για ένα σημαντικό άλμα στον καθορισμό μη στρατιωτικής πολιτικής. Ο κ. Αστρεβίτσιους το είπε άλλωστε καθαρά, αλλά βέβαια είναι ικανοποιημένο γι' αυτό, ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι εδώ ότι επιτέλους υπάρχει δυνατότητα ένα πρώην καθαρά πολιτικό, δηλαδή μη στρατιωτικό εργαλείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα και για στρατιωτικές επεμβάσεις. Ο κ. Ντανζόν στην τελευταία συζήτηση άλλωστε μας δήλωσε καθαρά ότι και στρατιωτικά νοσοκομεία είναι καθαρά ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ ότι εντάσσονται στο, στρατιωτικό ε, πλέγμα. Αυτά είναι ξεκάθαρα για την πλειοψηφία εδώ και τα χαιρετίζει. Όμως εγώ καθιστώ σαφές ότι εκτός του παρόντος σώματος αλλού στην κοινωνία των πολιτών, όπως για παράδειγμα και σε εκκλησιαστικές οργανώσεις οι οποίες συχνά συζητούν τέτοια θέματα, τα πράγματα αυτά δεν τα βλέπουν έτσι με μεγάλη φρίκη σημειώνουν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται και για στρατιωτικούς σκοπούς. Και σας επισημενω λάβετε υπόψη τις συζητήσεις αυτές που διεξάγονται στην κοινωνία και μην να αρκείστε να λέτε ότι πρόκειται μονάχα για τυπικότητες και για να ακολουθήσετε την οδό που υποδεικνύει ο εισηγητής. Δεν είναι πολιτικό, λέει δίθεν το θέμα, αλλά καθαρά τεχνικό. Εμείς πάντως ως Ενωτική Αριστερά είμαστε απολύτως αντίθετες με την εξέλιξη αυτή. Έχω καταθέσει και τροπολογίες και δεν στεκόμαστε απλώς κριτικά απέναντι στην πρόταση, την απορρίπτουμε. Έχω υποβάλει, όπως είπα, τροπολογίες που απηχούν αυτή την θέση. Για μας πρόκειται για κατάφορη κατάχρηση και αντιστροφή του χαρακτήρα των ε, διατάξεων αυτών. Θεωρώ λοιπόν ότι έρχονται σε απόλυτη αντίθεση και με τα δηλούμενα από το άρθρο 41 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του 208 όπου μιλούν για αναπτυξιακή βοήθεια και που πρωτίστως πρέπει να έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας. Ευχαριστώ πολύ. η εισηγήτρια των Πρασίνων, κυρία Βαλέο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας στην κυρία Λόζινγκ ότι αυτά τα οποία είπε δεν ήταν καθόλου βαρετά και πολλά από αυτά θα ήθελα να τα υποστηρίξω. Καταρχάς για τους πρασίνους είναι σαφές ότι έχουμε να, κάνει, να κάνουμε, αν θέλετε, με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ανάπτυξης βλέπει την υπόθεση αυτή. Και κατανοούμε ότι ο κύριος Ντονζόν θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, αν και οι αλλαγές αυτές ε, ε, σημειώνω ότι δεν είναι πάρα πολλές. Να πω ότι η νομική βάση για το συγκεκριμένο μέσο αυτό είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης και τεχνικής συνεργασίας με την βιώσιμη ανάπτυξη σαν στόχο. Όταν μιλάμε για την αναπτυξιακή πολιτική, ο κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Η ασφάλεια και η ανάπτυξη συμβαδίζουν, αλλά δεν ιεραρχούνται. Συνεπώς λοιπόν η εντύπωση από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι ότι η ασφάλεια είναι πιο σημαντική Πολλές φορές το αντίθετο είναι δυστυχώς πιο σημαντικό. Εμείς λοιπόν σαν πράσινοι έχουμε πιέσει για την χρήση του συγκεκριμένου μέσου και για περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της πρόληψης ε, των συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε επίπεδο συνεπειών στους αμάχους. Ε, δεν είναι ξεκάθαρο εδώ για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι, σαν παράδειγμα για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι στην ουσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και δυνατότητες οικονομικές από άλλους μηχανισμούς όπως το Αθηνά. Και εμείς έχουμε πει ότι τέτοιου είδους μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την ε, ε, Ένωση την Ευρωπαϊκή στον τομέα της ασφάλειας. Η ΚΕΠΑ, σαν παράδειγμα, θα μπορούσε να πάρει κάποιες αποφάσεις γύρω από αυτό. Επίσης δεν έχουμε κάνει τη σωστή διάκριση σχετικά με τον στρατιωτικό χαρακτήρα δράσεων και τον πολιτικό χαρακτήρα. Άμα πάρει κανείς τα χρήματα από την ανάπτυξη, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει σε τομείς οι οποίοι να είναι συμβατοί με τους στόχους του ΩΣΑ και αυτό όπως λέγεται θα πρέπει να είναι duckable με τα υπόλοιπα στοιχεία της οικονομικής μας παρέμβασης. Εκεί που όπως λέει το 3α, αυτά που λέει το 3α θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα κριτήρια DAC. Όπως είπε ο κύριος Ντονζόν, στην ουσία μιλάμε για έναν κανονισμό, δεν μιλάμε για μια έκθεση. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Και όταν βγάλει κανείς το exceptional με το specific και το αντικαταστήσει με το specific, το έκτακτο γίνεται εξειδικευμένο ή ειδικό. Το ειδικό μπορεί να είναι γενικής χρήσεως, ενώ το έκτακτο είναι μόνο έκτακτο. Συνεπώς το specific που χρησιμοποιείται δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς και χρήζει ε, περισσότερων διευκρινήσεων. Έχουμε εδώ μια διαφορετική αντίληψη από τον κύριο Τονζό. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει το κείμενο να εξασθενήσει, όπως το προτείνει ο κύριο Τονζό. Τώρα, ε, γιατί θα πρέπει να βγάλετε την ανάπτυξη από την τροπολογία 5. Η εξήγηση η οποία δίδεται δεν μας ικανοποιεί. Από ό,τι φαίνεται ο εισηγητής θεωρεί ότι η ασφάλεια είναι σημαντικότερη από την ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε όμως και για τα δύο μαζί, όχι για την ιεράρχησή τους. Συνεπώς λοιπόν η πολιτική μου ομάδα θα καταθέσει ορισμένες προτάσεις έτσι ώστε να υπογραμμίσει αυτά τα οποία είπα στην παρέμβασή μου και νομίζω ότι δεν θα σας εκπλήξει ε, το ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Περνάμε τώρα στον εισηγητή της ΔΕΒΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Βάιρινεν. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης και πρέπει να σας πω ότι ανησυχούν βαθύτατα και τα μέλη της Επιτροπής για τον κανονισμό αυτό. Υπάρχει ένας φόβος. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ε, των πόρων της αναπτυξιακής βοήθειας για ε, σκοπούς που δεν είναι πάντα οι προβλεπόμενοι από τον κανονισμό αυτό. Ε, που δεν γίνονται πάντα αποδεκτοί, ενώ οι προτεραιότητες μπορεί να βρίσκονται αλλού και θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια αυτά ε, για άλλους σκοπούς και μπορεί να είναι και εις βάρος της ποιότητας. Καλά μπορεί κάποιος να σου πει ότι είναι μικρό το ποσό, 25 εκατομμύρια μόνο, αλλά στο μέλλον ε, φοβόμαστε μήπως αυξηθεί και το ποσό αυτό και μήπως αλλάξει ριζικά η ίδια η φύση της αναπτυξιακής πολιτικής και χρηματοδότησής της. Διάφορες ήταν οι προτάσεις που συζητήθηκαν για το τι να κάνουμε. Κάποιος είπε ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει μια θέση του προπολογισμού ε, που να προέρχεται μόνο από την ΚΕΠΑ και να μην χρησιμοποιείται ε, προϋπολογισμός από την αναπτυξιακή βοήθεια θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση αυτή. βεβαίω ένα μέρος του ποσού να, πρέπει να αναφέρεται στον ΟΑΣΕ. Υπάρχει και μια γραμμή λοιπόν στον προπολογισμό της ΚΕΠΑ και εκτός αυτής τη χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιστώσεις τη αναπτυξιακή πολιτική για τη συνεργασία, το, το αντίστοιχο μέσο, την αναπτυξιακή συνεργασία και τον αντίστοιχο κανονισμό. Προσωπικά, ως εισηγητής, μάλλον συντάκτης γνωμοδότησης, δέχτηκα τη βασική ιδέα του κανονισμού, αλλά για να εξασφαλίσουμε και τους όχους της αναπτυξιακής πολιτικής στον λόγο κανονισμό, ε, πρότεινα να υπάρχει μία ρήτρα αποδοχής, accountability clause, δηλαδή να υπάρχουν κριτήρια το Φεβρουάριο του 2016 ε, είχαμε μια αναθεώρηση ε, του μέσου ODA για την, ε, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, δηλαδή για την ασφάλεια και την ειρήνη. Προτείνω μια τροπολογία επίσης που θα ενισχύσει τις αρχές και θα τονίσει τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής με βασικότερο στόχο την εκρίζωση της φτώχειας. Υπό την προϋπόθεση αυτή θα μπορούσε να δεχτεί έστω και με βαριά καρδιά η Επιτροπή ΔΕΒΕ Αναπτυξιακής Πολιτικής. Είναι πολύ νωρί για να πω τίποτα οριστικό γιατί δεν το έχουν συζητήσει οι σκιώδεις ηγητές. Έχω και κάποια προσωπικά σχόλια για ανησυχίε ω αναπληρωματικό μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε εξαιρετικέ περιστάσει και για συγκεκριμένου ε, σκοπού. Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής μας θέλει να αλλάξει τις εξαιρετικές περιστάσεις και να τις κάνει ειδικέ περιστάσεις που αποδυναμώνει. Και επίσης ε, διαγράφει τελείως τον όρο ανάπτυξη στην τροπολογία 5. Τον έφερε και η κυρία Βαλέρο προηγουμένως. Και ίσως το πιο δύσκολο σημείο να είναι το εξής. Ο συνδυασμός των τροπολογιών 7 και 8. Στην παράγραφο 3 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την εξής αρχή. Δηλαδή ε, ότι θα πρέπει να πληρούνται ε, όλες οι προϋποθέσεις ε, του α και β. Δηλαδή είναι συνολική ε, η ρύθμιση. Και στο σημείο α αναφέρει το όρος «και», το οποίο έγινε «ή», διαζευκτικό. Άρα θα πληρείται μόνο το β, όχι και το α και το β, οπότε θα είναι αρκετό. Αυτό είναι ριζική παρέμβαση και αλλαγή στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επιπλέον, στο σχέδιο έκθεσης, ναι, τελειώνεται λέει ο Πρόεδρος, συντομεύεται. Ναι, συντομεύω, τελειώνω. Ε, λοιπόν, ε, στο Β γίνεται λόγος για την διεθνή κοινότητα και Ή. Και αυτό έχει διαγραφεί. Λοιπόν, συμπέρασμα. Έχω την εντύπωση ότι το σχέδιο έκθεσης που συζητούμε θα ανοίξει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επεμβαίνουν στρατιωτικά στα θέματα ε, της άμυνας των ε, εταίρων τρίτων χωρών. Οι υπόλοιποι ομιλητέ, ο κύριο Γκάλερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Sorry. Um... Δεν ζήτησα το λόγο, λέει ο κύριο Γκάλερ. Καλώ. Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, ο κύριο Λίτ. Ε, ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ υπό διπλή ιδιότητα. Είμαι σκιώδης συγητής της Επιτροπής Αναπτύξεως και ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Κυρία Λόιζινγκ όχι, δεν ήταν βαρετά αυτά που είπατε. Τονίσατε πράγματα τα οποία συζητούμε και εμείς στην πολιτική μας ομάδα. Όχι αποκλειστικά, αλλά στο βασικό θέμα συμφωνούμε. Δηλαδή η εργαλειοθήκη της ανάπτυξης, τα χρήματα δηλαδή της αναπτυξιακής πολιτικής ασφαλώς και οφείλουν να εξυπηρετούν την αντιμετώπιση της φτώχειας. Συμφωνώ σε αυτά με τον εισηγητή. Δεν μπορεί να υπάρξει διαγραφή των κονδυλίων της αναπτυξιακής βοήθειας εν ώψη και των στόχων του 2030. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι ένα τέτοιο εργαλείο έχει αναπτυχθεί στην ε, Γερμανία 130 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Είναι σημαντική η προσέγγιση αυτή και σωστή. Έχει διπλό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, η γραμμή που ακολουθούμε στη Γερμανία μου φαίνεται σωστή και εδώ. Θα ζητήσουμε ως πολιτική ομάδα και εδώ να υπάρξει μια καθαρή γραμμή δεν σημαίνει ότι κονδύλια που δεν προέρχονται από τον προπολισμό για την ανάπτυξη πρέπει να περικοπούν. Αυτή είναι η γνωμοδότησή μας για την ώρα. Πρόεδρος, αν έχω καταλάβει καλά, ο κύριος Κέλαμ ζητάει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω με την ευκαιρία να υποστηρίξω την προεσέγγιση του συναδέλφου Ντανζάν ήμουν και παλαιότερα σκιώδης συγήτής του Λαϊκού Κόμματος για το Instrument for Stability. Σταθερότητας τότε τώρα είναι και ειρήνης. Η αφετηρία θα πρέπει να είναι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δηλαδή οι αλλαγές αυτές θα ενισχύσουν την διασύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Και είναι σαφές ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Λοιπόν, νομίζω ότι ο εισηγητής ξεκινά από αυτή την αντίληψη ότι δηλαδή η ασφάλεια έχει αμεληθεί, πάντως έχει ε, δυσχερανθεί η προσέγγιση σε αυτήν. Γι' αυτό και υποστηρίζω την ε, στάση του ε, στις τροπολογίες 2 και 3 που πρέπει να περιληφθεί ένα στοιχείο ευκαμψίας που δεν σημαίνει ότι δίνεται λευκή επιταγή για παρεμβάσεις σε τρίτες χώρες. Όμως αυτό το exceptional, αυτό το εξαιρετικό, να αντικατασταθεί από το αναγκαίο και εξειδικευμένο, τους όρους δηλαδή. Πρέπει να κατανοήσουμε και καλύτερα τι ακριβώς εννοεί. Διότι έχουμε 25 εκατομμύρια Πάντως είναι σημαντικό το εργαλείο αυτό για να προληφθούν και να σταθεροποιηθούν καταστάσεις στην άμεση γειτονία μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμφωνήσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να θεσπιστούν οι συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη στις τρίτες χώρες τις οποίες στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ της Επιτροπής αν επιθυμεί κάποιος εξημών να λάβει το λόγο, παρακαλώ να αυτοσυστηθείτε πρώτα. Θα μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον κύριο Νταονζόν για το σχέδιο εκθέσεως του, που νομίζω ότι προσφέρει γενική στήριξη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσεξε πολύ την σύνταξη της προτάσεως της, ώστε να διασφαλίσει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην συμπερίληψη ενός νέου παράγοντα, του στρατιωτικού παράγοντα δηλαδή, και την νομική βάση. Γι' αυτό δεν, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει το κέντρο βάρους της προσέγγισης για να ενταχθεί η προσπάθεια αυτή στην ΚΕΠΑ. Λέχθηκε και προηγουμένω ότι υπάρχει δυνατότητα να υπαρχθεί στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Αλλά θα είναι τότε πολύ διαφορετική η διαδικασία. Πολύ σύντομα τώρα, όσον αφορά τα θέματα που τέθηκε σχετικά με την DACability, με την δυνατότητα υπαγωγής στην ε, δράση της ε, Επιτροπής Αναπτυξιακής Στήριξης. Όπως είναι τώρα, δεν είναι ντάκαμπολ. Ένα μέρος των κονδυλίων μπορεί να δαπανηθεί, της και δηλαδή, και σε πράγματα τα οποία δεν υπάγονται στην ΤΑΚ. Όμως, 90% σχεδόν των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ICSP, είναι ντάκαμπολ και δηλώνεται ως τέτοιο εκ των υστέρων. Και δεν αναμένουμε η ισορροπία αυτή να αλλάξει πολύ, ακόμα και με τη νέα τροποποίηση. Να σας δώσω λίγα παραδείγματα. Μια τρέχουσα δραστηριότητα η οποία δεν υπάγεται στην DAC υπό το ICSP. Για να σας δώσω μια ιδέα περί τίνων δραστηριοτήτων μιλούμε. Υποστηρίζουμε για την ώρα την αποστολή ΟΑΣΕ στην Ουκρανία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Μίνσκ ή την αποτυχία εφαρμογής της Συμφωνίας Μίνσκ. Δεν πρόκειται για στήριξη της ανάπτυξης της Ουκρανίας. Πρόκειται για στήριξη στην Συμφωνία του Μίνσκ. Γι' αυτό και δεν θεωρούμε την ε, δαπάνη αυτή τα καμπολ. αλλά είναι μια αναγκαία στήριξη για να μπορούν να λειτουργήσουν οι παρατηρητές επιτόπου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από την ICSP, δεν είναι duckable, αλλά θεωρούμε ζωτική σημασία και ότι εντάσσεται στα πλαίσια του εργαλείου αυτού όσο έχει σήμερα. Σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη του στρατού στην εφαρμογή της προτάσεως στο μέλλον, αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι πλαίσια τα οποία είναι έκτακτα, όπως στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με φορείς εξωτερικών δράσεων που και με, με, φορείς ε, τόπου, όπως η αστυνομία και η χωροφυλακή στη χώρα αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι οι στρατιωτικοί φορείς μέσα σε τέτοια πλαίσια δεν είναι σε διαφορετική κατάσταση από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν ενδεχομένω χάσει την δυνατότητα επέμβαση για την προστασία του πληθυσμού και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και απειλή κατά του πληθυσμού. Το ίδιο όπως θα μπορούσαν να είναι και μέσω προστασίας του. Άρα πολλά από τα μέτρα που θα αναλάβουμε να επιβάλλουμε με τη βοήθεια του στρατού είναι για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Έχουμε δηλαδή περιστάσεις, για παράδειγμα, ε, ενώ και πάλι την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου υπάρχουν στρατώνες, όπου σημαίνουν τα επιθαρχία μεταξύ των στρατιωτών. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ανοιχτοί οι στρατώνες και μπαινοβγαίνει κόσμος. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό με κάποιο στοχευμένο τρόπο. Η πρόταση αυτή θα μας επιτρέψει από την άποψη της ανάπτυξης να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε ώστε να μείνουν οι στρατιώτες στους στρατώνες και τα όπλα να είναι ασφαλή όσο δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του στρατού. Τέτοιου είδου δραστηριότητε δηλαδή θεωρούμε ότι οι ορισμένε περιστάσεις τέτοια μέτρα ασφαλείας είναι σημαντικά πριν να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί η ειρήνη. E e e? Ευχαριστώ. Από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θέλει κανεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από πλευρά μα δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε απολύτω τα όσα είπε ο συνάδελφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια μικρή αναφορά μόνο στο εξή γεγονό. αν θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί επαναστατικό βήμα. Εγώ θα ήμουν πιο μετρημένος σε εκφράσεις, ότι είναι και αυτό κάτι που εντάσσεται στην παρούσα τάση, ε, όπου συνδυάζεται η ασφάλεια με την ανάπτυξη, είναι πιο στενά συνδεδεμένες. Έγινε αναφορά κατά τη διάρκεια της συζήτησης στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το 16. Συνδέονται λοιπόν περισσότερο, όλο και περισσότερο αυτές οι δύο έννοιες και αυτή είναι η βάση για τη σημερινή πρόταση και τη συζήτηση. Για τα υπόλοιπα με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής θέλει να επανέλθει, κύριος Ευχαριστώ, έγιναν παρεμβάσεις ε, τις οποίες έχουμε ήδη ακούσει μέχρι τώρα στη συζήτηση. Να υπενθυμίσω γενικά ότι εγώ ναι μεν κατανοώ αυτό που λέγουν ορισμένοι συνάδελφοι, ότι εμείς είμαστε υπέρ της σύνδεση της ασφάλειας με την ανάπτυξη, φιλοσοφικό. Αλλά όταν μιλάμε για την πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου δεσμού, για το τι θα κάνουμε με αυτό το κείμενο, το οποίο είπα είναι μετριοπαθέστατο, ε, επανερχόμεθα στις αρχικές ιδεολογικές θέσεις που λέγουν ότι κοιτάξτε αν συνδέσουμε την ανάπτυξη με την ασφάλεια, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι ισχυρότερη της ε, ανάπτυξης. Ας θυμίσουμε λίγο εδώ την τάξη μεγέθους. Οι με μεγέθους για την ΚΕΠΑ για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός λοιπόν, ο τακτικός 13-20 είναι 31 δις. Ε, δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα τα οποία είναι περιορισμένα, προσθετικά και τα οποία δεν απορφούν πιστώσεις από αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν κινήσει σε διαφορετικά επίπεδα. Είναι συμπληρώματα πολιτικών και προγραμμάτων. Συνεπώς λοιπόν ε, είναι λίγο εύκολο να αποδίδει κανείς προθέσεις για ένα μέσο το οποίο ε, είναι πλήρες, αυτόνομο, χρηματοδοτούμενο αυτονόμος επίσης και που δεν δημιουργεί προβλήματα και ανισορροπίες. Ε, πού τις βλέπετε εσείς τις ανισορροπίες σας αυτές ανάμεσα στα χρήματα που δίδονται για την ανάπτυξη από τη μία στον προϋπολογισμό. Τώρα για το DACABLE, το συμβατό με το DAC. Κοιτάξτε, είναι νομίζω λάθος ε, ε, η, η εξίσωση αυτή. Ακριβώς γίνεται μία προσπάθεια για να μην έχουμε ε, ένα πρόγραμμα το οποίο να μην είναι DACABLE. Δεν θα πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε με λάθος τρόπο το συγκεκριμένο μέσο. Ένα άλλο σημείο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι κάνω ρητορική για να αποφύγουμε την πολιτική συζήτηση. Ε, δεν θα πρέπει να γράψουμε μια έκθεση μέσα στην οποία θα βάλουμε όλες μας τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές απόψεις και θα εγκαταλείψουμε έναν κανονισμό που θα έπρεπε αντίθετα να γίνει αποτελεσματικότερος. Και μου λέτε να βγω από το κοινοβούλιο και να ε, ανοιχνεύσω τις απόψεις των μεν και των δε. Κοιτάξτε, εγώ έχω επαφή και με έξω και με το εσωτερικό του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι αυτά τα οποία προτείνουμε δεν τα ζητούν τα βιομηχανικά και στρατιωτικά λόμπι. Ας πούμε, οι αρχές του Μαλή, οι οποίες χάνουν έναν στρατιώτη την ημέρα και μας λένε ότι δεν έχουμε ε, κλινικές εκστρατείας, νοσοκομεία εκστρατείας με τόπου. Συνεπώς λοιπόν ότι στα μέσα Ιανουαρίου υπήρξαν 80 νεκροί και 150 τραυματίες στον ΚΑΟ. Φυσικά οι αρχές του Μαλή και οι υπηρεσίες που είχαν δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες και τα νοσοκομεία τα στρατιωτικά των Γάλλων κυρίως, αλλά όχι μόνο, ήταν αυτοί που έκαναν τη δουλειά και φρόντισαν τους τραυματίες. Λοιπόν, δεν κάνω ασκέτη ρητορική, στήρα ρητορική. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να δούμε πού χρησιμεύουν τα χρήματα αυτά και να είμαστε συγκεκριμένοι. Όταν μας λέγουν ότι οι αποστολές μας και πά, ε, στην ουσία καταρτίζουν αλλά δεν δίδουν ε, εξοπλισμούς στρατιωτικούς. Φυσικά δεν δίνουμε τάγκ εμείς, δεν δίνουμε τεθωρακισμένα στον στρατό της Κέντρο Αφρικανικής Δημοκρατίας. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες που έχουν οι στρατιώτες, οι μαχητές, οι επίσημοι και η ανάπτυξή τους στο μέτωπο είναι κάτι στο οποίο το κάνουν με πάρα πολύ καλό τρόπο και με μεγάλη χαρά οι Τούρκοι, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε σε δημοσιονομικό και σε νομικό επίπεδο και να το κάνουμε και εμείς. Έλαβα επίσης υπόψη κάποιες άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τις τροπολογίες. Θα ε, προτείνω στους Κιώδης να τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες διατυπώσεις επακριβέστερες, αυστηρότερες, πιο συγκεκριμένες μάλλον, που να ανταποκρίνονται στις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει για ένα κείμενο που είναι κανονισμός. Είναι νομικός κανονισμός και δεν είναι μια οδηγία ή μια έκθεση που θα επέτρεπε την ευρύτερη και γενικότερη έκφρασή μας γύρω από ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους ομιλητές. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι η προθεσμία κατά απολογιών 8 Μαΐου στις 11 λέει ο Πρόεδρος. 26 Ιουνίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή ενώ στις, στις 11 Ιουλίου θα τελειώσω και θα επανέλθουμε. 11 Ιουλίου και μετά θα πάει στην Ολομέλεια. Ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν σήκωσα φαίνεται αρκετά ψηλά την κάρτα μου, λέει ο κύριο Κάρβερ. Σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριο Ντανζάν. Δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι θέλουμε να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό μας έχουν κλέξει όλους εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκπαιδεύει ε, στρατιωτικούς. Τα κράτη-μέλη διμερώς τα κοιτούν αυτά. Έχει όλο και περισσότερες ε, στρατιωτικές φιλοδοξίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς. Σέβομαι και τα επιχειρήματα που ακούω, αλλά η διατύπωση έχει προσοχή. Λέτε ότι τα έχουμε κοιτάξει προσεκτικά και τα διατυπώνουμε προσεκτικά. Τα είπε και η κυρία Λόζεν και άλλοι συνάδελφοι. το θέμα είναι πάρα πολύ ε, αφιλεγόμενο ε, και στη διατύπωση. Είναι πάρα πολύ αμφίσιμη η διατύπωση για τη δράση τη στρατιωτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο επιλέγουμε αυτές τις διατυπώσεις. Συμπεριλαμβάνονται και άλλες οργανώσεις ασφαλείας, ακόμα κάποια μισθοφορικά σώματα σε όλα αυτά. Το 42.2 γίνεται λόγος για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση με εξαίρεση ε, κάποια στρατιωτικά και αμυντικά ζητήματα όπου η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μάλλον εκτός αν έχει αποφασίσει ομόφωνα το Συμβούλιο. Ακόμα και αν λέτε ότι υπάρχει τέτοια επιχείρηση είναι πολύ αφιλεγόμενη διατύπωση και αφήσιμη. Κοιτάξτε, δεν θα ξανανοίξουμε τώρα τη συζήτηση, θα τα κοιτάξουμε αυτά και θα φροντίσουμε ε, στις ε, νεδράσεις των σχεδόν ε, εισηγητών να συμμετέχει και η ομάδα σας, η ευθυντή. Λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ το σημείο 6 με τις ανακοινώσεις που σας έκανα και θα προχωρήσουμε στο σημείο παριθμών 7 και 8 σε κοινή συζήτηση. Έχουν φτάσει οι ομιλητές μας, οπότε θα τους παρακαλέσουμε να έρθουν στο Προεδρείο. Okay. So... Λοιπόν, συνεχίζουμε το σημείο 7 και 8 από κοινού, όπως είπαμε. Ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ. Φιλοξενούμε δύο εμπειρογνώμονες σήμερα στην Επιτροπή μας. Πρώτος είναι ο κύριος Κάιβερς, διευθυντής του Κέντρου Σπουδών ΑΣΕΑΝ στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και μετά θα γίνει συζήτηση για τις πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΑΣΕΑΝ. Θα εορτάσει την 50η επέτειο της φέτος η ΑΣΕΑΝ και έχουμε και την 40η επέτειο των επισήμων σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ είναι εταίροι ως ε, βασική περιφερειακή παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΑΣΕΑΝ. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αναβάθμιση των σχέσεών μας σε στρατηγικό επίπεδο και τον Ιούλιο του 2014 επιβεβαιώθηκε από την Υπουργική Συνάντηση αυτή. Το 2015 η Πατή Εκπρόσωπος ενέκρινε μια κοινή ανακοίνωση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΑΣΕΑΝ μια εταιρική σχέση με στρατηγικούς στόχους». Εκεί έχουμε έναν οδικό χάρτη λοιπόν ε, που εμβαθύνει τη συνεργασία μας σε επίπεδο πολιτικής συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής δραστηριότητας φυσικών πόρων. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Κέπερς για 10 λεπτά και ελπίζω να έρθει και ο συναδελφός σας, ο έτερος εμπειρογνώμος σε λίγο. Um, Κυρίες και κύριοι, στο παρελθόν Υπήρξαν κάποιες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ ε, λόγω του λεγόμενου ασιατικού τρόπου λειτουργίας εντός εισαγωγικών. Το 1967 άρχισε να λειτουργεί επίσημα και στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70 στόχος ήταν η πολιτική συνεργασία μεταξύ των μελών ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασφαλείας. Τότε στόχος δεν ήταν ακόμα η περιφερειακή ολοκλήρωση. Οι χώρες έβγαιναν από την απεικιοκρατία και η ανεξαρτησία τους οδήγησε σε αντιπαλότητες, σε και κάποια προβλήματα μεταξύ τους. Άρα για το λόγο αυτό έγινε κάποια θεσμική συνεργασία που σήμερα είναι γνωστή ως ε, Asian Way. Αυτός ο ε, τρόπος λειτουργίας όμως εμποδίζει τις μελλοντικές εξελίξεις και τις θεσμικές δομές συνεργασίας. Ο Asian Way ως τρόπος ε, των προβλημάτων εδράζεται σε κάποιες κοινότητες της Μαλαισίας που ε, με διαβουλεύσεις ε, ε, συμμετείχαν στη λύση διαφόρων προβλημάτων. Υπάρχει μια ευελιξία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν στην εργασία τους και στην περιφερειακή ολοκλήρωση όσο το επιθυμούν. Όχι περισσότερο. Οι αποφάσεις εντός της ΑΣΕΑΝ λαμβάνονται κυρίως συνενετικά. Και θέματα που δεν μπορούν να λύσουν μεταξύ τους οι χώρες συχνά το βάζουν στην άκρη για να μην επηρεάζουν τη συνεργασία σε άλλους τομείς. Γι' αυτός ο τρόπος λειτουργίας ΑΣΕΑΝ εντός εισαγωγικών συχνά έχει επικριθεί ε, ως χρονοβόρος, αργός και λίγο παραγωγικό στην οικονομική ολοκλήρωση και με σκαμπανεβάσματα στις συμφωνίες, ε, τις εμπορικές ε, ελευθέρων συναλλαγών που είχαμε στη δεκαετία του 90. Πιο πρόσφατα έχουμε και άλλα παραδείγματα, μεταξύ αυτών την εφαρμογή της συμφωνίας για την ε, οικονομική κοινότητα ΑΣΕΑΝ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να τονίσουμε το εξής. Ουδέποτε είχαν σκεφτεί τελωνιακή ένωση και οικονομολόγοι εξέχοντες ΑΣΕΑΝ πάντα προειδοποιούν κατά της Θελωνιακής Ένωσης Για παραθέτω εδώ ότι δεν είναι αριστικό μοντέλο για την συνεργασία μεταξύ χωρών ΑΣΕΑΝ. Μια τελωνιακή ένωση θα σημαίνει εκχώρηση σημαντικών ε, εξουσιών και αρμοδιοτήτων ε, ε, εθνικής αρμοδιότητας σε ένα υπερεθνικό επίπεδο που είναι πολιτικά ανέφικτο γιατί αντιτίθεται στην μέθοδο με την οποία λειτουργεί ο ΣΕΑΝ, αλλά και δεν είναι και βιώσιμη αυτή από οικονομικής πλευράς, γιατί θα σήμαινε μια κοινή εμπορική πολιτική, εξωτερική πολιτική σε χώρες μη μέλη τη ΑΣΕΑΝ και πιο περιοριστική από αυτοί που ακολουθούν κάποιες μεγάλες χώρες μέλη της ΑΣΕΑΝ όπως είναι η Σιγκαπούρη. Μετά τη δημιουργία του χώρου ελευθέρων συναλλαγών του 2002 στην ΑΣΕΑΝ, οι χώρες μέλη το 2007 έκαναν μια σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε μέχρι τα τέλη του 2015 να δημιουργηθεί μια οικονομική κοινότητα ως ένας από τους τρεις πυλώνες της ΑΣΕΑΝ. Αλλά ε, η προθεσμία 2015 ξέπνευσε χωρίς να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και θεωρήθηκε ως ορόσημο απλώς προόδου παρά καταλεκτική ε, χρονιά παραμένουν πολλοί φραγμοί και εμπόδια μη τελωνιακού χαρακτήρα και το χρησιμοποιούν αυτό κατά τη γνώμη μου ως δικαιολογία κάποιες χώρες ΑΣΕΑΝ για να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για το τι για... γιατί συμβαίνει αυτό. Κυρίως επειδή δεν υπάρχουν ε, θεσμοί σε επίπεδο ΑΣΕΑΝ που να υποστηρίζουν την ολοκλήρωση, που και αυτό με τη σειρά του ε, οφείλεται στην αποστροφή που έχουν οι χώρες μέλη της ΑΣΕΑΝ για μια ε, συγκεντρωτική μορφή συνεργασίας ε, πολιτικής και δεν πρόκειται να αλλάξει στο προσεχές μέλλον αυτή η νοοτροπία. Ένα άλλο σημαντικό είναι οι τεράστιες διαφορές στην ανάπτυξή τους Υπάρχει ένα χάσμα περιφερειακό ανάπτυξη τη ΑΣΕΑΝ. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό μεταξύ των χωρών μελών. επίγον είναι να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα σε επίπεδο ΑΣΕΑΝ. Αλλά αυτό δεν το αναγνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες χώρες με ε, ικανοποιητικό τρόπο. οι συγγραφείς διανοούμενοι και ε, πανεπιστημιακοί των χωρών αυτών που γνωρίζουν το δόγμα που λέγεται Asian Way ε, Λένε ότι είναι τέσσερις ε, χώρες που είναι πιο ανεπτυγμένες, η ε, ε, Βυρμανία, το Βιετνάμ, που αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από τις υπόλοιπες έξι, CLMV. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη σύγκληση και αναμένεται μεγαλύτερη σύγκληση. Βέβαια, απομένει να αποδειχθεί αν η σύγκληση αυτή θα γίνει με αρκετά ταχύ ρυθμό. Μέχρι το 2013 έχει υπολογιστεί ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Σιγκαπούρη σε σύγκριση με την Καμπότζη Φερρυπίν ε, ήταν 59,8 φορές μεγαλύτερο τη Σιγκαπούρη στο ΑΕΠ από την Καμπότζη. και αναμένεται μέχρι το 2030 αυτός ο λόγος, αυτό το κλάσμα που είναι 59,8 να έχει γίνει 27. Ε, τολμώ να αμφιβάλλω αν αυτό είναι ε, αρκετό για να υπάρξει σύγκληση στο μέλλον. Πέραν λοιπόν από την αξιοπιστία και από το γεγονός ε, ότι εξαρτώνται οι χώρες αυτές από ε, τις υποδομές και τους διαδρόμους υποπεριφερειακούς μαζί με την ε, τράπεζα ε, την αναπτυξιακή της Ασίας, η ΑΣΕΑΝ έχει δημιουργήσει σημαντικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα. Όπως είναι η πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση ΑΣΕΑΝ με τις προτιμησιακές σχέσεις που έχουν οι έξι χώρες προς τις χώρες CNV που είναι Καμπότζη, Λάος, ε, Μίανμαρ και Βιετνάμ. Υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν περιφερειακής συνεργασίας ε, που θα βοηθήσουν τις χώρες που το χρειάζονται περισσότερο να πλησιάσουν τις πιο αναπτυγμένες. Η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να εστιάζεται ε, στην ε, ανάπτυξη, στην κατάρτιση εργαζομένων, στην απόκτηση δεξιοτήτων για την ανταγωνιστικότητα. Και οι χώρες ΑΣΕΑΝ συνεισφέρουν όσο μπορούν η καθεμία εντό αγωγικών και παράθεση αυτό που δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχει γίνει αναφορά στο πλαίσιο αυτό στα ταμεία συνοχής και στα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, χωρίς να αντιστοιχεί απολύτως. Ε, και είναι και πολύ παραπλανητική αυτή η σύγκριση. Αν δείτε τι συμβαίνει εκεί. Η πρωτοβουλία AIA από την αρχή, από το σχεδιασμό της, κυρίως κινείται ε, από ε, τη Μαλαισία και την ε, Σιγκαπούρη ε, με τα, βάσει τα δικά του συμφέροντα και μοντέλα. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες θετικής διάκρισης των χωρών CLMV, ταυτόχρονα έμεσα και άμεσα αναγνωρίζεται ότι όλα τα μέλη, όλα τα μέλη θα πρέπει να υποφελούνται από τη συνεργασία. Σε κάποιο βαθμό αυτό συμβαίνει, καταβάλλονται προσπάθειες για να ε, ολοκληρωθεί η κοινότητα ΑΣΕΑΝ, αλλά το πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι δεν γίνεται, δεν δίνεται μεγάλη προσοχή σε πραγματικές περιφερειακές πολιτικές στην ΑΣΕΑ ή σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης και ε, υπάρχει ένα χάσμα, επαναλαμβάνω, μεταξύ των κρατών ΑΣΕΑΝ. όπως είναι οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, στο εσωτερικό των κρατών αυτών υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Βεβαίως, μεταξύ των χωρών ΑΣΕΑΝ, δύο μόνο έχουν καθεστώς υψηλού εισοδήματος. Άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της περιοχής από την ίδια την ΑΣΕΑΝ ή από τις τέσσερις χώρες Καμπότζη, Λάος, ε, Βερμανία και Βιετνάμ. Και αναπτυξιακή τους βοήθεια συχνά θεωρείται κάτι που στρέφεται κατά του εθνικού συμφέροντος και ενίσχυση μελλοντικών ανταγωνιστών. Οπότε δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ε, ε, τη ρητορική που ακούμε για μείωση ε, των διαφορών και του χάσματος δεν γίνονται συγκεκριμένα βήματα για να μειωθεί όντω αυτό το χάσμα. Και όταν γίνονται είναι αναποτελεσματικά. Και από επίπεδο, ξέρω εγώ, πολιτικής οικονομίας μπορεί κανείς κοινικά να περιγράψει την τρέχουσα κατάσταση ως κυρίαρχη λύση ενός παιχνιδιού συντονισμού. Αυτά τα ξέρουν και τα περιγράφουν έτσι οι οικονομικοί επιστήμονες. Και πάλι με τον ασιατικό τρόπο λειτουργίας της ΑΣΕΑΝ, με συνενετικό τρόπο λήψης αποφάσεων, αργό και αναποτελεσματικό. Και από τη μία έχουμε τις έξι χώρες ΑΣΕΑΝ, από την άλλη CLM, τις χώρες 4 CLMV και τους δωρητές σε ένα διεθνές περιβάλλον και περιφερειακό που αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρουν ένα τρόπο να αντιμετωπίσουν ε, το χάσμα, το αναπτυξιακό, να ασχοληθούν με τα έργα ε, με ε, την πρόθεση της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό είναι ένα έργο που αναλογεί στη γραμματεία ΣΕΑΝ. Αλλά ε, οι χώρες αυτές δεν το δέχονται. Δεν δέχονται να πάρουν πρωτοβουλίες τα σώματα αυτά, οι θεσμοί όπως είναι η γραμματεία ΣΕΑΝ, χωρίς να έχουν συμφωνήσει προηγουμένως οι χώρες μέλη για να αυξηθεί ε, η δράση και να χειραφετηθεί η λειτουργία σαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε και τον δεύτερο ε, ομιλητή μας σήμερα, τον κύριο Ντέιλι της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων και αρμόδιο για θέματα ASEAN. Ευχαριστώ να ακούσουμε την τοποθέτησή σας. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μας ως Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και για το πώς επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίθετο. Γνωρίζω ότι συζητείτε σήμερα σχέδιο εκθέσεως για το ζήτημα αυτό, κάτι που αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντός σας το οποίο εκτιμά ιδιαίτερα η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Φέτος είναι σημαντικό έτος, διότι μεταξύ άλλων είναι και η 40η επέτειος της ενάρξεως του διαλόγου και σχέσεων μεταξύ ΑΣΕΑΝ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντικός υποστηρικτής της περιφερειακής ολοκλήρωση της Νοτιοανατολικής Ασίας για λόγους ανάπτυξης και σταθερότητας. Οι ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασιαν είναι πολύ σημαντικές για μας. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρος για την ολοκλήρωση αυτή είναι μοναδικού χαρακτήρα εταίρος για την περιοχή αυτή του κόσμου, διότι εμείς κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες ΑΣΕΑΝ για την περιφερειακή ολοκλήρωση. Και ανεξαρτήτως των λεπτομεριών των προκλήσεων αυτών που τόσο εύγλωτα εξήγησε ο κύριος καθηγητής, παρόλα αυτά η Ένωση ως Ένωση μπορεί να πει ειλικρινώς στους, στις χώρες αν κοιτάξτε είμαστε πραγματικά μοναδικός εταίρος για σας γιατί κατανοούμε ακριβώς το, ποιο είναι το, το, το, το εγχείρημα. Υπάρχουν ε, περισσότερες επισκέψεις υψηλού επίπεδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ειδικό ε, πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2015 για σχέση με το ΑΣΕΑΝ συνεχίζονται οι διαδικασίες και η συνεργασία δεσμευόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των περιοχών αυτών του κόσμου που εκπροσωπούμε εμεί και η ΑΣΕΑΝ η 21η συνάντηση ε, υπουργών που έγινε τον Οκτώβριο πέρσι επιβεβαίωσε ότι είναι πιο διαθρωμένες και πιο ισχυρές οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ των δύο πιο προχωρημένων διαδικασιών ολοκληρώσεως στον κόσμο εξακολουθούν να παραμένουν πολύ σημαντικές και ιδίως τώρα σε μια εποχή ε, παγκόσμιας αστάθειας η στρατηγική σχέση που να βασίζεται σε συγκεκριμένα υλοποιήσιμα αποτελέσματα μεταξύ ΑΣΕΑΝ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το βάθεμα των σχέσεών μας και το να γίνουν πιο φιλόδοξες αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα υπέρ του σκοπού αυτού με την εφαρμογή των αποφάσεων της συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών που λήφθηκαν το 2014 και επαναλήφθηκαν πέρσι. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχωρούν σε διάφορους τομείς. Οι διαπραγματεύσει για μια σε βάθος συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές προχωρούν καλά. Και αναμένουμε ο τρίτος γύρος να διεξαχθεί τούτο το μήνα στο Ελσίνκι. Οι Υπουργοί Οικονομικών ΑΣΕΑΝ μαζί με τον δικό μας Ευρωπαίο Επίτροπο συναντήθηκαν τον Μάρτιο στην Μανίλα των Φιλιππινών για την τρίτη συνάντηση και για διαβουλεύσεις οικονομικού χαρακτήρα. Σημειώσαμε τις σημαντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που ανέρχονται σε 208 δισεκατομμύρια αξίας ευρώ. Πέρσι δηλαδή πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάθε δύο ημέρες. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάθε δύο ημέρες. Ξαναλέω, είμαστε ο δεύτερος σημαντικότερος εταίρος της ΑΣΕΑΝ και ο ΑΣΕΑΝ ως συνασπισμός είναι ο τρίτος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μάλστρομ, Ευρωπαία Επίτροπος για το Εμπόριο, σε συνεργασία με τους υπουργού ε, των χωρών ΑΣΕΑΝ, προχωρούν για τη σύναψη συμφωνίας ε, ελεύθερου εμπορίου. Λίγα λόγια για την συνεργασία για την ασφάλεια τώρα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί σε στενότερη συνεργασία με τις χώρες ΑΣΙΑΝ για την ασφάλεια και άμυνα. Σημαντική δέσμευση, η οποία θα συνεχιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά διακυβεύματα στην ασφάλεια της περιοχής αυτής, δηλαδή έχει πολλά πράγματα που την ενδιαφέρουν και οι χώρες αυτές αντλούν από τη δική μας εμπειρία. Μεταξύ των πρωτοβουλειών που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη φέτος είναι και ένα σεμινάριο ERF για την ανακοπή των εξτρεμιστικών τάσεων που έγινε στις Βρυξέλλες. Φέτος επίσης για τη διακίνηση ή μεταφορά προσώπων ένα orientation course που, που γίνεται μάλλον στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα και ένα σεμινάριο ERF για ζητήματα συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης, στην Μιανμάρ αυτό, στα τέλη Ιουνίου. Η τέταρτη ε, διαδικασία διαλόγου υψηλού επίπεδου θα γίνει το δεύτερο εξάμεινο φέτος στις Φιλιππίνες. Ως μέρος αυτής της αναβάθμισης των σχέσεών μας και για να ανταποκριθούμε σε φωνές που ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ένωσης στην περιοχή αυτού του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει στην αναβάθμιση των, ε, της ατζέντα σημαντικών οργανώσεων όπως τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΑΣΕΑΝ. Υπάρχει μια λογική βάση σε αυτό, διότι πιστεύουμε στην εξέλιξη της ΑΣΕΑΝ και στον ε, συγκεντρωτικό της χαρακτήρα, διότι πιστεύουμε στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΑΣΕΑΝ. Γι' αυτό για μας ως λογικό συμπέρασμα είναι αναγκαίο να παίξουμε ένα σημαντικότερο ρόλο σε όλα τα φόρουμ όπου ηγείται η κίνηση ΑΣΕΑΝ. Επί της ουσίας, σε όλους τους τομείς προτεραιότητας αυτοί συμβαδίζουν και με τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, συμμετέχει, ε, ήδη διαθέτει σημαντική ε, εμπειρία, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του διεθνούς, της διεθνούς εγκληματικότητας, για την διαμεσολάβηση και ούτω καθεξής. Και όπως έχουμε αποδείξει, και, στα, και στο ε, Περιφερειακό Φόρουμ ΑΣΕΑΝ. Γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κοινή κατανόηση ότι ΑΣΕΑΝ και Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία ήδη διαθέτει σταθερά θεμέλια. Σε τέτοια συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία, θα πρέπει να συμβάλλουμε μεν στην στήριξη των δε πιο ενστικτοδός και να συζητούμε ζητήματα παγκόσμιας ισχύω, ξεπερνώντας το καθαρά διμερές επίπεδο. Θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο ρόλο παίζουμε σε διαφορετικά ε, διεθνή φόρουμ, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στη Γενέβη, είτε αλλού. Κύριε Πρόεδρε, ειδού λίγα λόγια που ήθελα να σας απευθύνω για να θέσω το πλαίσιο των ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Αυτό το οποίο θα κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να συνδυάσουμε τα δύο σημεία. Καταρχάς θα δούμε ποιοι σκιώδεις είναι διαθέσιμοι. Βλέπω τον εισηγητή. Δεν είμαι τόσο μικρός όμως, λέω. Κύριος Μπουτιχόφερ. Λοιπόν, συγγνώμη, θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή λοιπόν για να μας παρουσιάσει την δική του πρόταση και να θέσει ερωτήσεις στους δύο εμπειρογνώμονες και μετά θα επανέλθουμε μετά από το γύρο των ερωτήσεων. Κύριε Μπουτιχόφερ, έχετε το λόγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και τους δύο εμπειρογνώμονες. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ελπίζω για να υπογραμμίσω κάποια από τα σημεία τα οποία πιστεύω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην έκθεσή μου, την οποία όλοι έχετε στη διάθεσή σας. Καταρχάς θα ήθελα σε επίπεδο διαδικασίας να πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η αύριο 12 το μεσημέρι. Η εξέταση στην ΑΦΕΤ προβλέπεται στις 19 Ιουνίου, η ψηφοφορία στις 20 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον μήνα Σεπτέμβριο. Έμαθα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι η κυρία Μογκερίνη θα ταξιδέψει στην περιοχή τον μήνα Αύγουστο και ίσως να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς της εξωτερικής δράσης να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την έκθεσή μας η οποία να έχει ήδη ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο στην ανακοίνωση την οποία θα κάνουν στην περιοχή. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δούμε αν τεχνικά αυτό είναι εφικτό να διοργανώσουμε διαφορετικά τη χρονική εξέλιξη, να ψηφίσουμε τον Ιούλιο και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την άποψη του Κοινοβουλίου μαζί με αυτή της εξωτερικής δράσης. Τώρα να έρθω στην ουσία. Λίγα πράγματα να υπογραμμίσω, να πω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να θέτει κανείς στόχους για την ΑΣΕΑΝ και για την ανάπτυξή τους σαν περιφερειακό σώμα γιατί δεν είναι ρόλος μας. Ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για την περιφερειακή ολοκλήρωση και να υποστηρίξουμε επίσης και την πολιτική που λέγει ότι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κεντρικό χαρακτήρα της ΑΣΕΑΝ. Νομίζω επίσης ότι και αναφέρομαι εδώ στο άρθρο 5, στην παράγραφο 5 μάλλον, της πρότασης ψηφίσματος, πιστεύω ότι έχουμε την δυνατότητα να ασκήσουμε αυτοκριτική εν μέρη, διότι στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή συνάντησα πολλούς οι οποίοι άσκησαν κριτική για την ασθενική στάση την οποία είχαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όπως η διαφοροποίηση ε, για τα θέματα των νήσων της νότιας συνικής θάλασσας. Θα πρέπει λοιπόν και με τις ενέργειές μας και όχι μόνο θεωρητικά να αντιδράσουμε γύρω από αυτό το θέμα. Ε, πιστεύω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς πιστεύαμε στο παρελθόν. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταστεί ένας αξιόλογος εταίρος για μη συμβατικές ανησυχίες στον τομέα της ασφάλειας για πάρα πολλά θέματα. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό σαν ε, δυνατότητα. Η παράγραφος 8 αναφέρονται επίσης και στην ε, Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορικών Σχέσεων. Είχα μία συνάντηση με τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, η οποία πιστεύει ότι η διατύπωση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ισχωρούμε, ότι παρεμβαίνουμε σε ευθύνες της Επιτροπής ΣΥΝΤΕ, θα προτείνω κάποιες αλλαγές, αλλά επί της ουσίας όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυξημένο για μια συμφωνία με την περιοχή και γι' αυτό θα πρέπει να μην την αγνοήσουμε. Και γι' αυτό είχα και συνάντηση με την κυρία Μάλστομ, η οποία συμφωνεί με τους στόχους που έχουμε θέσει. Δύο επιπλέον σύντομα σημεία. Φέτος έχουμε, θα έλεγα, γενέθλια πολλά και για μας και για την ΑΣΕΑΝ. Είχα πολλούς συνομιλητές για την ιδέα να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία ε, για μια ανταλλαγή προγραμμάτων, για ένα πρόγραμμα μάλλον ανταλλαγών νέων ηγετών από την Ένωση και από την ΑΣΕΑΝ για να γιορτάσουμε τα γενέθλια των ΜΕΝ και των ΔΕ και να χαράξουμε ένα νέο δρόμο για το μέλλον. Εγώ έχω πάρει θετικές αντιδράσεις από αρκετούς ομιλητές εδώ, ε, εμπλεκόμενους και στις Βρυξέλλες και στην περιοχή και μπορούμε να το προωθήσουμε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή. Τέλος, ε, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα να δώσουν προτεραιότητα σε υψηλή συχνότητα πολιτικών επαφών. Ο μοναδικός τρόπος για μας να μπορέσουμε πράγματι να τύχουμε πλήρους αναγνώρισης ως αξιόπιστος εταίρος, ως πολύτιμος εταίρος στο μέλλον για το ΑΣΕΑΝ, είναι να μην χάνουμε τις ευκαιρίες τις οποίες έχουμε για συνεργασία πλήρως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούτιχόφερ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούτιχόφερ Συμφωνώ με την αντίληψή του για την έκθεση αυτή. Δεν θα επαναλάβω τα θετικά στοιχεία τα οποία είπε ήδη. Ελπίζω η έκθεση αυτή να ξεκινήσει, να οδηγήσει στο να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση ωφέλιμη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μορφές συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση και τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Σχετικά τώρα με τον λεγόμενο ασιατικό τρόπο ή τον τρόπο ΑΣΕΑΝ, εμείς θα πρέπει να στηρίζουμε την ολοκλήρωση την περιφερειακή που θα οδηγήσει ίσως σε μια ενιαία αγορά και σε περαιτέρω επαφές ανάμεσα σε ε, πρόσωπα κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ασφάλεια στην περιοχή. Νομίζω ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μας με μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου είναι ζωτική συνεργασία στην έρευνα, στην καινοτομία, την εκπαίδευση, τη συνδεσιμότητα είναι θέματα που πρέπει να ενισχυθούν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διμερείς ελεύθερες συμφωνίες σαν θεμέλια για μια ευρύτερη συμφωνία εμπορική. Πολλές φορές θεωρούμε ότι οι σχέσεις μας με την ΑΣΕΑΝ είναι αυστηρά οικονομικές ή εμπορικές, ενώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάρε πέραν αυτής της αντίληψης οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ μπορεί να αναυξηθούν ακόμα περισσότερο Συμφωνώ με τη στρατηγική συνεργασία με την περιοχή. Είναι κομβικό για τις μελλοντικές σχέσεις μας να έχουμε πιο ισχυρές πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Και εδώ υπάρχει δυνητικά και κάποιος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον διακοινοβουλευτικό διάλογο και την συνεργασία με την διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕΑΝ. Έχουμε πολύ συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα υπόλοιπα περιφερειακά σώματα. Μπορούμε λοιπόν να αναστρέψουμε την προσοχή μας στην ενίσχυση και ανάπτυξη των σχέσεων αυτών. Ευχαριστώ τους δύο εμπειρογνώμονες για τις δηλώσεις τους. Ήταν χρήσιμες οι δηλώσεις τους, ήταν ε, πραγματικά υποβοηθητικές της προσπάθειάς μας. Ένα σχόλιο να κάνουν παρακαλώ. Η ολοκλήρωση ΑΣΕΑΝ έχει φτάσει τα 50 πια χρόνια. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς και οικονομικά και πολιτικά. Έχουν ε, βέβαια οι χώρες ΑΣΕΑΝ την δυνατότητα να συνεχίσουν την εμπειρία αυτή, αλλά θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε και εμπειρίες ε, με τη δική μας περιφερειακή εμπειρογνωμοσύνη. Ο κύριος Κιουτσούκ, χωρίς μικρόφωνο. Ο κύριος Μποστινάρου, θέλω να μιλήσω εγώ εξ του δικού μας κοιόδου. Α, δεν ε, σα ξέχασα την ομάδα σας, αλλά δεν ξέραμε ποιο θα μιλήσει από εσά. Ωραία, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω εξ ονόματο του συναδέλφου David Μάρτιν. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεση του κύριου Μάρτιν. Το 2017 έχουμε την 40η επέτειο των σχέσεών μας με την ΑΣΕΑΝ και τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό και να στραφούμε προς το μέλλον. Έχουμε πλέον ε, ισχυρούς οικονομικούς ε, δεσμούς που θα πρέπει να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε με δύο ε, συμφωνίες που ερημένουν την υπογραφή τους και σταματώ εδώ με τις στατιστικές. Δεν είναι μόνο οικονομικός εταίρος σημαντικός αλλά και στρατηγικός, περιφερειακός για την ασφάλεια και την σταθερότητα. Ιδιαίτερα ε, ε, όταν επικρατεί τέτοια βεβαιότητα και αστάθεια παγκοσμίω. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει παρουσία εκεί. Κοιτάξτε τι αποφασίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, για το πώς θα τοποθετηθούν στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένωση αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατικών δικαιωμάτων. Εργασιακών αυτά είναι σημαντικά για μας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα θέτουμε υπόψη των συναδέλφων ε, και στο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άρχισε το 2015 και καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τις Εμπορικές. Για να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή ΑΣΕΑΝ θα πρέπει να έχει στόχο να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Που οι πολίτες τώρα ζητούν ε, ελεύθερο τύπο, ε, μεγαλύτερες ελευθερίες για τις αναδυόμενες μεσαίες τάξεις. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μειονότητα των Ροχίνγκια στην Βερμανία, Μίανμαρ ε, και στην Ταϊλάνδη, στη Μαλαισία, την Ινδονησία και αλλού έχουμε προβλήματα, χιλιάδες εκτελέσεις εκτός δίκης στις Φιλιππίνες με περιορισμό των ελευθεριών ε, έκφρασης, των ελευθεριών ε, του ε, συνεταιρίζεστε σε διάφορες χώρες έχουν δει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να παραμένουν ατιμόρυτες. Αν θέλει η να αναπτυχθεί, να έχει αξιοπιστία και να αναγνωρίζεται ως ένας παγκόσμιος στρατηγικός εταίρος και παίκτης για την ασφάλεια της περιοχής, για την ασφάλεια, τη θαλάσσια και το εμπορίο. Ευχαριστώ ξερώματος του David Μάρτιν. Εγώ σε ευχαριστώ. Και τώρα η φιλελευθέρη. Η ΣΥΑΡ δεν θα μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κόφερ για τι προσπάθειες του, λέει ο για την εκπόνηση τη έκθεση αυτή για τι πολιτικέ μα σχέσει με την ε, ΑΣΕΑΝ. Είναι συνολικές, καλύπτουν πολλούς τομείς και το εμπόριο και τι επενδύσει και την ανάπτυξη και τα πολιτικά ζητήματα. Είναι πολύ επίκαιρη η έκθεση αυτή γιατί γιορτάζουμε την 40η επέτειο των επισήμων σχέσεών μα. Είναι από τις πιο δυναμικές ε, περιφέρειες του κόσμου, αυτή που καλύπτει η ΑΣΕΑΝ, με ταχύτητα τους ρυθμούς ανάπτυξης και θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη σχέση μας. Δεν θα πρέπει αυτό να το παραβλέψουμε. Το Δεκέμβριο του 2014 δώσαμε στις Φιλιππίνες το καθεστώς των ε, εμπορικών προτιμησιακών σχέσεων. GSP+, και αυτό θα πρέπει να είναι έμπνευση και για τις υπόλοιπες χώρες. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει ε, η σχέση μας να αναβαθμιστεί, να γίνει στρατηγική σχέση, είναι σπουδαία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Ασία. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε στην έκθεση και την ανησυχία μας για τη διάβρωση της δημοκρατίας, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την συνεχιζόμενη καταπίεση και τις διακρίσεις σε διάφορες χώρες, ιδιαίτερα στις Φιλιππίνες και στη Μιανμάρ, Ιρμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόχμπίλερ, τελευταία ομιλήτρια των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητρία γιατί βέβαια δικός μας είναι ο βασικός συγητής. Έχω όμως ερωτήσεις προς τους ομιλητές, καθώς και μια ερώτηση προς τον εισηγητή, κύριο Μπιουτικόφερ. Περιλαμβάνεται πολλές διατυπώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην έκθεση και σωστά. Ως κανόνα δεν ξεχωρίζουμε χώρες για να τις κατονομάσουμε. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όμως έτσι, διότι στην Μιανμάρ και στις Φιλιππίνες βλέπουμε σημαντική οπισθοδρόμηση στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να μην τα αναφέρουμε φαίνεται παράξενο. Για τους ομιλητές τώρα, ερώτηση προς τον κύριο Κάουβαρτ. Λέτε ότι δεν βλέπετε πολύ πραγματική συνεργασία μεταξύ των ίδιων των χώρων μελών ΑΣΕΑΝ. Τι έχετε να πείτε για αυτή την υποπεριφερειακή συνεργασία σε ορισμένες περιοχές του κάτω Μεκόγκ για παράδειγμα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Ίσως έχετε και άλλα παραδείγματα όπου μια τέτοια συνεργασία δεν απέδωσε. Για τον κύριο Ντάλι, είπατε ότι αυτά τα 50 χρόνια συνεργασίας των ΑΣΕΑΝ πρέπει να στηριχτεί μπορείτε να είστε κάπως πιο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Μποστινάρου είπε ότι έχουμε έναν διάλογο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ ήδη από την πρώτη συνάντηση του 2015. Προβλέπονται περισσότερα πράγματα σχετικά στο προσεχές μέλλον. Ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ενδιαφέρον για μια πολιτική στενότερης διασύνδεσης μεταξύ ευρωπαϊκών, ε, ε, εμπορικών σχέσεων με ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, Φιλιππίνες που έχει τώρα ε, καθεστώς GSP συν και έχουμε όμως μπορεί ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ξεκινήσει η διαδικασία κατά του Προέδρου της χώρας αυτής. Η συνεργασία αυτή, για παράδειγμα και στην επιστήμη, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση αντί σε επιδείνωση της καταστάσεως. Και τέλος επίσης, κύριε Ντάλη, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΑΣΕΑΝ θα πρέπει να συνεργαστούν συνολικά και σε πολλά επίπεδα. Αλλά για ποια θέματα. Για θέματα μετανάστευσης εν ώψη και των ε, χωρών συνεργασίας του Περισσικού Κόλπου, βλέπω εκεί ότι άλλες χώρες έχουν ε, ε, κάποιες θετικές πολιτικές. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος. Ευχαριστώ, λέω, Προεδρεύων. Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, ως συνήθως. Ας απαντήσουν οι δύο εμπειρογνώμονες, αν μπορείτε να το κάνετε όμως σε δυόμιση λεπτά ο καθένας. Φιλόδοξο μεν, αλλά θα είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χρόνου της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω λίγα λόγια για την περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον. Θα ήθελα να πω γι' αυτό δύο πράγματα ή να αναπτύξω λίγο περισσότερα. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών. Νομίζω ότι η πολιτική προσέγγιση είναι σωστή. Δηλαδή, όταν κατέστη σαφέ ότι την εποχή εκείνη δεν ήταν δυνατό ε, να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των δύο την εποχη εκεινη δεν ηταν δυνατο να γινουν διαπραγματεύσει μεταξυ των δυο περιφερειων να προτιμηθεί η εθνική προσέγγιση, δηλαδή να ε, γίνει διαπραγμάτευση συμφωνίας με Σιγκαπούρη, Βιετνάμ κλπ. Πάντως για έναν αριθμό λόγων, ένας από τους οποίους λόγους ήταν ότι η ΑΣΕΑΝ ομάδα χωρών δεν συγκρίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έχει κεντρικό θεσμικό χαρακτήρα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο, όπως είπα πριν, είναι η μεγάλη αναπτυξιακή απόκληση μεταξύ των χωρών ΑΣΕΑΝ. Ορισμένες χώρες μάλιστα είναι και διστακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις αυτές. Όμως γνωρίζετε ήδη ότι ορισμένες αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΣΕΑΝ, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαπραγματεύεται με τι χώρε μέλη τη άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα πράγμα που ήθελα να πω. Το δεύτερο ε, έχει σχέση με την διαφορά, με την απόκληση στην ανάπτυξη. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Οι χώρες αυτές χρειάζονται πολύ βοήθεια και νομίζω ότι με την χορήγηση περισσότερη στήριξη στις λιγότερο ή και στις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες ΑΣΕΑΝ θα τους επιτρέψουμε να λειτουργήσουν καλύτερα, να ενταχθούν καλύτερα στην ΑΣΕΑΝ και επομένω θα τις βοηθήσουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δική μας σκοπιά. Τέλος για τη συνεργασία στον Μεκόγκ. Έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι τόσο επιτυχημένη η συνεργασία αυτή. Πάντως προωθείται δημόσια ως πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Δεν είναι όμως και τόσο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πάντως μία από τις λίγες περιφερειακές συνεργασίες που ε, έχουν επιτύχει σε έναν βαθμό. Αρχικά η συνεργασία άρχισε υπό την αιγίδα της ε, Asian Development Bank και σε κάποιο βαθμό που άρχισε να επιτυγχάνει, άρχισε να μπαίνει στα επίσημα έγγραφα ASEAN σαν, να ήθελαν με τον τρόπο αυτό να προσελκύσουν τη δημοσιότητα και να ε, προχωρήσουν σε μια ε, πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι όντως είναι κάτι το σημαντικό. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά που ετέθησαν τα ερωτήματα πρώτα για την ολοκλήρωση της ΑΣΕΑΝ μετά από 50 χρόνια, πώς μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί διακαώς να μοιραστεί την εμπειρία της με άλλες περιφέρειες ε, του κόσμου και τώρα στην ΑΣΕΑΝ. Βέβαια δεν μπορεί να μεταφερθεί ένα προς ένα η εμπειρία. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και συζητήσεις εξηγούμε πώς έχουμε φτάσει σε κάποια επιτεύγματα, πώς προχωρούμε, πώς δρούμε και σε ποιες περιπτώσεις οι χώρες εάν μπορούν να θεωρήσουν χρήσιμο και ωφέλιμο κάποια από τα δικά μας ε, επιτεύγματα για να αντιμετωπίσουν δικές τους προκλήσεις και προβλήματα. Και αυτό είναι η κεντρική ιδέα σε όλους τους ε, διαλόγους και τους τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαμε διάλογο με την Επιτροπή, ΑΣΕΑΝ, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΑΣΕΑΝ και τους επόμενους μήνες επίκειται και άλλη μια τέτοια συνεδρίαση. Βεβαίως, εκτός των διμερών διαλόγων που έχουμε με, με τις μεμονωμένες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρονται η κατάσταση στην Ταϊλάνδη, το θέμα των Ροχίνγκια, το θέμα των Φιλιππινών επίσης όλα αυτά μας ανησυχούν και θέτουμε τις ανησυχίες μας υπόψη των χωρών αυτών στις άμεσες επαφές που έχουμε μαζί τους. Ε, για το DSGP+, στον κανονισμό προβλέπεται αυτό το σύστημα προσημεκών σχέσεων για να ενθαρρύνουμε τις χώρες να αρθούν στο ύψος ε, διεθνών συμβάσεων με σημαντικό περιεχόμενο, θέματα εργασιακά, περιβαλλοντικά, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν μια χώρα λαμβάνει τέτοιο καθεστώς, υπάρχει και ένα ε, ολόκληρο σύνολο, μια δέσμη επιτήρησης ή παρακολούθησης των δράσεων. Και στις Φιλιππίνες η αποστολή μας μετέβει φέτο, στι αρχές του έτους και βρισκόμαστε σε επαφή και σε συνεργασία. Τα παγκόσμια ζητήματα, ποια είναι αυτά. Πώ ορίζονται. Συνήθως θέματα όπως η κλιματική αλλαγή ή θέματα ασφαλείας μας επιβάλλονται ως παγκόσμια ή καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εκτός από τη μετανάστευση. Και το θέμα που μας ενδιαφέρει μας και το θέτουμε όπως και άλλοι, ε, στη συνεργασία μας και την αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες ΑΖΕΑΝ, εμείς θέλουμε να μπούμε στην ουσία των θεμάτων ε, σε περιφερειακό επίπεδο, πέρα από το αμυγός διμερές και να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οικονομικός αλλά και πολιτικός εταίρος και δεν ενδιαφέρεται μόνο για ζητήματα διμερούς ε, ενδιαφέροντος με τη στενή έννοια, αλλά με την ευρεία και την παγκόσμια έννοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συγητής ζήτησε να επανέλθει. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους σε σχέση με την ερώτηση που μου έκανε η κυρία Λόχ Μπίλερ. Δεν θεωρώ όντω ότι είναι δική μου ευθύνη στην παρούσα έκθεση να κατονομάζω ε, συγκεκριμένες χώρες. Έχουμε ψηφίσματα για το σκοπό αυτό ε, στο Κοινοβούλιο. Στις αιτιολογικές αναφορές αναφέρω τουλάχιστον 11 ε, ψηφίσματα, οπότε καλύπτουμε το έδαφος αυτό στη συνέχεια. Με όλο το σεβασμό διαφωνώ με την επιφύλαξη του κυρίου Κέρβερς για ε, τον στόχο να συνεχίσουμε και να ε, αποσκοπούμε σε μια περιφερειακή ε, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και υπάρχουν και προσδοκίες από την περιφέρεια που προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πάει ευκαιρία αυτή χαμένη. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Για το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να απαντήσω σε ερωτήσει του, προ... του προλήσαντος Στην Επιτροπή μας θα γνωμοδοτήσουμε θα δώσουμε μάλλον την έκθεσή μας και θα τα λάβει υπόψη αυτά η πατή εκπρόσωπος ε, και ενδεχομένως αν χρειαστεί να έχουμε και τα αποτελέσματα της δικής της επίσκεψης ε, για την Ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ΙΝΤΑ, ε, θα κάνουν τροπολογίες. Ε, αν δεν μπορούν να το κάνουν για λόγους χρονικούς, ε, ο δικός μας σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι ο μόνιμος εισηγητής της ΙΝΤΑ για την ΑΣΕΑΝ και μπορεί να το λάβει υπόψη και να τα εντάξουμε και στη δική μας έκθεση. Και φυσικά δεν μπορούμε να, να μην έχουμε καμία απολύτως αναφορά στο ελεύθερο εμπόριο στη δική μα έκθεση, επειδή δεν είμαστε ίντα. Αυτά. Τα τεχνικά λοιπόν τώρα που έχω να σας πω. Αύριο λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες στις 11 λέει ο, ο μιλητής. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η πρωινή μας συνεδρίαση. Ραντεβού στις 3, όπου έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στις 3 η ώρα.